Uh, Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα σας παρακαλούσα όλους να καθίσετε. Νομίζω ότι αρκούν οι θέσεις για τους ε, επισκέπτες μας. Να καλωσορίσω θερμά τους ε, συμμετέχοντες ε, στην ε, στρογγυλή τράπεζα που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα που έχει οργανωθεί από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που έχει θέμα την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη ελληνική αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Έχει οργανωθεί η στρογγυλή τράπεζα αυτή από την εισηγήτρια για μια σημαντική έκθεση πρωτοβουλίας μας, την Άννα Μαρία Κοράτσα την οποία καλωσορίζω θέρμα. Ε, θα με βοηθήσει στον συντονισμό των διαδικασιών σήμερα και ε, χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω ε, ε, μια σειρά διακεκριμένων προσκεκλημένων. Λογικά έχετε έναν κατάλογο όλων των ομιλητών. Έχετε και πρόγραμμα. Οπότε έχετε κανονικά ένα φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι παρόντες πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι. Βλέπω πολλά γνωστά πρόσωπα στο κοινό. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια στρογγυλή τράπεζα. Δεν είναι επίσημη ακρόαση του Κοινοβουλίου και ξέρω ότι οι βουλευτές συνάδελφοι θα θέλουν να ε, συμμετάσχουν στη συζήτηση. Θα θέλαμε όμως στο στάδιο αυτό να ακούσουμε ε, ομιλητές και από το κοινό. Για να το κάνουμε αυτό σας ε, έχουμε δώσει ένα έντυπο εγγραφή, εάν θέλετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση ή εάν ε, ήρθατε εδώ με σκοπό να πείτε κάτι πολύ σημαντικό μπορείτε να ε, συμπληρώσετε το έντυπο ε, θα υπάρχουν άτομα στην αίθουσα που θα συλλέγουν τα έντυπα μπορείτε να μας πείτε ποιος είστε, ποια οργάνωση εκπροσωπείτε και ως άτομα, ως μεμονωμένοι πολίτες αν είσαστε παρόντες και πάλι θέλαμε να ακούσουμε τη θέση σας. Είναι κάπως ε, πείραμα η σημερινή ε, στρογγυλή τράπεζα. Θα δούμε πώς θα, πώς θα πάει. Αυτά όσον αφορά τα τυπικά. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Εγώ ως ε, πρόεδρος θα παρακολουθώ το ρολόι ώστε να βοηθήσω όλους τους διακεκριμένους ομιλητές μας να τηρούν το χρόνο τους ώστε να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Να σας δώσω το πλαίσιο της εστρογγυλής αυτής της τράπεζας, τι ακριβώς ε, θέλουμε να πετύχουμε. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια που μαζί με τους κοιόδης εισηγητές, τους οποίους επίσης καλωσορίζω, είναι υπεύθυνοι για την ε, σημερινή ε, διοργάνωση. Άννα Μαρία, παρακαλώ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, Ένα λόγο που θα ε, είναι επιτυχή σημερινή συζήτηση είναι ότι ο Μάρκον Χάρμπορ δεν είναι μόνο πρόεδρος τη ΙΜΚΟ, είναι και σκιώδη συζητή μου και αυτό είναι πολύ καλό. Είχαμε ήδη πολύ καλό διάλογο και με του άλλου σκιώδης συζητητές και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Και ο άλλο λόγο είναι ότι η επιχειρηματική κοινότητα, ο τομέα τη Ελληνική έχει πάρει πολύ στα σοβαρά την έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας που βρίσκεστε εδώ, που ε, έχουμε συναντηθεί σε, ε, με διάφορους τρόπους το, το, το τελευταίο τρίμηνο, μεμονωμένα, διμερώς ή σε, σε επιτροπές. Ε, το όνειρό μου ήταν να έχω μια ζωντανή έκθεση και βλέπω να πραγματοποιείται το όνειρο, αυτό. Ε, ε, βλέπω να πραγματοποιείται ε, επικοδομητικός διάλογος. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον ε, Επίτροπο Παρνιέ, να, να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο Μπαρνιέ για την, για, για, για την βίβλο, για την λιανική ελληνική αγορά. Ε, να καλωσορίσω και τον κύριο Πελζοβάν για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, με ε, τη μελέτη του που αποτελεί τη βάση για τη δουλειά μας. Ε, μαζί με του συναδέλφου, μου έχουμε εντοπίσει τέσσερι βασικού τομεί, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν πρόκειται για μια νέα έκθεση ΒΟΒΕ, ούτε οδηγία για τα δικαιώματα των καναλατών ή για την επισήμανση. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι για να ε, έχουμε ε, αποτελέσματα θα πρέπει να ε, περιοριστούμε σε κάποια θέματα, να επικεντρωθούμε σε κάποια θέματα. Ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε με συγκεκριμένα παραδείγματα των προβλημάτων που συναντάτε στις καθημερινές εργασίες σας και να μας δώσετε Συγκεκριμένε προτάσει λύσεων για το τι μπορεί να γίνει από το Κοινοβούλιο, από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη για να λύσουμε τα προβλήματά σας. Και στο κάτω-κάτω αυτό που κάνουμε μαζί είναι ότι βοηθάμε να δημιουργηθούν θέσεις εργασία. Η έκθεσή μου έχει να κάνει με την απασχόληση. Ελπίζω μερικοί από εσά να συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι και να δούμε το φως στην άκρη του τούνελ ε, μετά από την ε, οικονομική κρίση, την ε, κρίση της ανεργίας, την κοινωνική κρίση ε, όλοι μας έχουμε κοινή ευθύνη ώστε να ε, έχουμε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για μένα η, θέση η απασχόληση βρίσκεται στο, ε, στο, στο, επίκεντρο, στο κέντρο της έκθεσής μου. Θέλουμε να ο καταναλωτής να έχει επιλογές και, να, και περισσότερη προστιθέμενη αξία. Για το λόγο αυτό δεν είδα τον ε, λόγο να χωρίσω την ε, έκθεση σε ε, κεφάλαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Eurocommerce και για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που πέτυχαν από μόνοι τους συμφωνία και που μας παρουσίασαν Ποιο πιστεύουν ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν ε, κάποια από τα προβλήματα της απασχόλησης στον τομέα. Για παράδειγμα, η ε, καταπολέμηση του, ε, του, του ανεπίσημου τομέα της μαύρης αγοράς. Επίσης, θα ήθελα να Ευχαριστώ να συμπεριλάβω κάποια από τα όσα θα υποθούν στην έκθεση. Να σας περιγράψω το όραμά μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε την πραγματική οικονομία στο, στην καρδιά της ε, πολιτικής ε, συζήτησης. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο χώρο στην ηλιανική αγορά. Οι καλές πρακτικές και η θετική συμβολή στην ε, δουλειά, στην, στην ζωή πολλών πολιτών θα πρέπει να τονιστούν. Ταυτόχρονα υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Το να αρνηθούμε την ύπαρξη των προβλημάτων δεν ωφελεί κανέναν. Υπάρχουν προβλήματα ε, ανάμεσα στους μεγάλους και τους μικρούς ε, λιανοπολιτές. Υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα, ε, μεταξύ των μεγάλων, υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ, γενικά σε όλο το μήκος της αλυσίδας διανομής. Μερικά από τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το δικαίωμα εγκατάστασης, τα μερίδια αγοράς, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ απέναντι στα κέντρα των πόλεων, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Ε, έχουμε το θέμα των εμπορικών πρακτικών, ε, των εμπορικών σχέσεων. Ελπίζω σήμερα πραγματικά να μπορέσουμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα. Νομίζω ότι η βασική μας πρόκληση είναι να ξεφύγουμε από την ε, σύγκρουση, από την άρνηση των προβλημάτων, από την απελπισία και να προχωρήσουμε σε έναν πιο επικοδομητικό διάλογο. Ο διάλογος πιστεύω θα πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα και ε, χαίρομαι που σήμερα θα ακούσουμε κάποια ε, γεγονότα. Ε, νομίζω ότι και άλλοι θα έχουν να μας παρουσιάσουν ε, γεγονότα. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδεολογία και από τους μύθους ε, και να προχωρήσουμε στα γεγονότα. Τι, ποιες είναι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, πώς τις ορίζουμε, υπάρχουν πραγματικά θα ήθελα να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Τι πιστεύετε σχετικά με το σύστημα πληρωμών στην ε, Ευρώπη. Θέλουμε να περικόψουμε τις, ε, το, το κόστος. Ε, οι τιμές είναι ο μόνος τρόπος να καθορίσουμε τι επιφέρει προστιθέμενη αξία για τους πολίτες. Θα ήθελα να ε, κλείσω εδώ τη δική μου ε, εισαγωγή, διότι είναι δική σας ημέρα. Θα ήθελα να ακούσω και τους συναδέλφους ε, και εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Μαρία, για την ενεργητική ηγετική σου στάση και εισαγωγή. Ας προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη συνεδρία. Έχετε το πρόγραμμα ενωπιών σας, επομένως δεν χρειάζεται να αναφερθώ στις διαφορές συνεδρίες. Έχουμε την πρώτη συζήτηση για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Εγώ λίγο θα πρέπει να μιλάω, έτσι λοιπόν αυτό είναι ενθαρρυντικό. Έχουμε τους δύο αρχικούς ομιλητές, ο Λουκ Χέντριξ είναι ο πρώτος, ο οποίος είναι διευθυντής για την αντιγωνιστικά των επιχειρήσεων της εξωτερικής σχέσης και νομικές υποθέσεις για τη UEAPMI, την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και ο Ξαβιέ ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του Eurocommerce και είναι η οργάνωση που εκπροσωπεί πολλές οργανώσεις λιανικής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν θα δώσω στον καθένα πέντε λεπτά και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Χέντριξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Κοράτσα. Αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ για την ε, πρωτοβουλία της να οργανώσει αυτή την ακρόαση για έναν πολύ σημαντικό τομέα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε που δίνετε και στη ΓΟΕΑΠ με τη δυνατότητα να συμβάλλει στη συζήτηση θα ήθελα να απαντήσω αρνητικά στις, ε, με αρνητικό τρόπο σε ερωτήσεις σας. Δηλαδή να σας πω ποιες, τι είδους νομοθεσία δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην ε, εσωτερική αγορά. Για την ΕΕ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Τι είδους λιανική αγορά θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας διαβάσει την έκθεση της Επιτροπής, ε, μένουμε με ένα αίσθημα σκεπτικισμού, διότι πολύ λίγη προσοχή δίδεται στους ε, μικρούς ανεξάρτητους λιανοπολιτές ε, και πολύ συχνά παρουσιάζονται αρνητικά. Τι σημαίνει πιο αποτελεσματική λιανική αγορά. Εάν αποτελεσματικότητα σημαίνει πιο αποδοτική, που είναι ο συνήθις οικονομικός ορισμός, τότε η Κομισιόν από την αρχή έδειξε προτίμηση για μορφές λιανικής με την υψηλότερη απόδοση. Με άλλα λόγια, με, ε, τον υψηλότερο τζίρο ανα, ε, ε, αναεργαζόμενο, δηλαδή προτίμηση για τους μεγάλους ελιανοπολιτές πέρα από τον παράγοντα οικονομία κλίμακας μπορεί να είναι σαφές ότι δεν είναι ο ο, πιο αποτελεσματικός, η, πιο ο πιο αποδοτικός τύπος αυτός. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν θέλει καταστήματα με λιγότερους ε, υπαλλήλους. Ε, μια ε, ε, λιανική αγορά που λειτουργεί καλά δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Η ΟΕΑΠΜΕ θέλει καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περισσότερη εναρμόνιση. Εναρμόνιση όμως δεν σημαίνει καθόλου ρύθμιση κατά τη γνώμη μας. Ε, δεν μπορούν να πετύχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς να διασφαλίσουμε την διόρθωση της ελεύθερης αγοράς και να υπάρχει ισορροπία και δυνατότητα για κάθε παράγοντα στην αγορά, μεγάλο ή μικρό, να έχει τις ίδιες ε, ευκαιρίες. Και ακριβώς αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ζητούν κάποιοι ακόμα, να, ε, να, εξαλειφθεί, να καταργηθεί η εθνική νομοθεσία που διασφαλίζει ε, ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους ε, τους παράγοντες της λιανικής αγοράς, μεγάλους και μικρούς. Κατά τη γνώμη της ΟΕΑΠ, με μια πραγματική εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, θα διασφαλίζει ένα ε, πλαίσιο με μεγάλη ποικιλότητα στο οποίο ο καταναλωτής ε, να ε, έχει ελεύθερη επιλογή ανάμεσα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και μικρά τοπικά καταστήματα. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα την απαγόρευση των πωλήσεων κάτω του κόστους. Αυτός, το, να επιτρέπουμε τέτοιες πωλήσει δεν σημαίνει μόνο ότι δεχόμαστε τον νόμο της ζούγκλας. Το δικαστήριο έχει επανειλημμένα ε, δεχτεί τη δυνατότητα να διατηρηθεί η απαγόρευση αυτή. Η ε, απαγόρευση αυτή είναι απαραίτητη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον λιανικό τομέα και δεν υπάρχει κανένα, ε, καμία απόδειξη ότι δεν είναι αποτελεσματική η σχετική νομοθεσία. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι κανόνες σχετικά με την... είναι οι κανόνες χωροταξίας. Το Σημαντικό είναι να υπάρχουν καταστήματα στα οποία να έχουν πρόσβαση και οι πιο ηλικιωμένοι. Η οδηγία περί υπηρεσιών ε, δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οικονομικά κριτήρια σχετικά με, την, ε, με το άνοιγμα καταστημάτων και ιδιαίτερα ε, σούπερ μάρκετ. Είναι όμως σαφές ότι κάποιοι λόγοι γενικού ενδιαφέροντος όπως είναι και ε, το περιβάλλον, ε, το αστικό περιβάλλον ε, κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των κανόνων για το άνοιγμα τέτοιων καταστημάτων λιανικής. Η ΟΕΑΠ επίσης πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική λιανικής θα πρέπει να σέβεται τα τις αρχές ε, της επικουρικότητας ε, και της αναλογικότητας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές λιανικής είναι απλά τοπικές αγορές. Σύμφωνα με την ΟΕΑΠΜΕ, ε, η Κομισιόν στην έκθεσή τη υπερτιμάει τη σημασία του διασυνοριακού εμπορίου και δεν είναι αυτή η απάντηση για να έχουμε μια λιανική αγορά με ποικιλότητα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών μια προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις διαφορετικές συνθήκες σε, στα διάφορα κράτη-μέλη και πολλά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, και ε, μια τέτοια προσέγγιση έχει, το περισσότερα πλεονεκτήματα από την ε, λεγόμενη εξάλληψη όλων των εμποδίων ε, στις εθνικές αγορές. Για παράδειγμα, οι ώρες καταστημάτων είναι ένα από τα θέματα που καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο κρατών μελών. Εάν θέλουμε να το ρυθμίσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε ε, πιθανότατα να υπάρχουν ε, λιγότερα εμπόδια για τους μεγάλους, ε, αλλά δεν καλύπτουμε έτσι τις τοπικές ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και που τηρήσατε και το χρόνο. Κατόπιν ο κύριος Ξαβιαντηρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι εξωτιμοί βουλευτέ, καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω με ευγνωμοσύνη μου στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ ε, για το ανοιχτό τη πνεύμα και την προθυμία τη να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα για να πετύχει μία αγορά για το εμπόριο προ όφελο των καταναλωτών και μάλιστα είδαμε ότι έγινε πριν προσπάθεια και πριν δύο εβδομάδες εγώ θέλω να σας πω ότι εκπροσωπώ 30 μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και 6 εκατομμύρια ε, για ε, μέσω της Ένωσης αλλά και χονδρέμπορους και επίσης ε, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη σήμερα το πρωί στο δικό μας Συμβούλιο. Εκτιμούμε ε, τη βούληση Επιτροπής και Κοινοβουλίου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα και αναγνωρίζεται στην έκθεση παρακολούθησης της αγοράς η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία και στην ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά. Ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο οδηγεί σε υψηλά ωφέλη για την ενιαία αγορά, κυρίως για τον καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός επιφέρει ποικιλία, ποιότητα, καινοτομία, φορεία στον καταναλωτή και αυτό συμβαίνει επιβάλλοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευαστικές ε, πέραν από τις νομικές απαιτήσει. Ε, ο Άλμπερτ Χάιν, ο οποίος επιβίωσε την περισμένη εβδομάδα, είπε ότι εμείς ε, δεν πολλούμε εκ μέρου του προμηθευτή, αλλά αγοράζουμε εκ μέρου του καταναλωτή. Η αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το ότι ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια. Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 2008 για να έχουμε μια δεσμή δεσμή μέτρων, η όπω ε, ήταν η οδηγία για τις υπηρεσίε. Και σήμερα εξακολουθούμε να βλέπουμε πολλές ελλείψεις στην εφαρμογή τη. Όμω αυτό το νομοθέτημα ε, ουσιαστικά μειώνει τον αυξανόμενο προστατευτισμό. Παρ' όλα αυτά, πολλά πρέπει να γίνουν για την άρση των εμποδίων και για τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών για καλύτερες τιμές και με μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογή των καταναλωτών. Μου ζητήσατε να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα και θα αναφερθώ σε ορισμένα είδη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε για προϊόν ή με κατασκευαστή και έχουμε κάποια παραδείγματα που προέρχονται από τον ίδιο τον επιχειρηματικό τομέα. Το πρώτο παράδειγμα έχει να κάνει με τον έλεγχο και την επιθεώρηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έγγραφα που έχουν να κάνουν με το προϊόν για την πώληση σε ό,τι αφορά και την αξιολόγηση ε, τη ε, ποιότητα και τη καναλότητα, θα πρέπει να τα έχει στην κατοχή του αυτό που θέτει πρώτο το προϊόν σε εμπορία. Στην πραγματικότητα, πολλά κράτη-μέλη ζητούν αυτά τα έγγραφα να είναι αμέσω διαθέσιμα σε επίπεδο λιανεμπόρου και πολλέ φορέ σε επίπεδο καταστήματο. Δεύτερο παράδειγμα είναι κάποια τεχνικά εμπόδια παρά το ότι η οδηγία του 98 αποτελεί, απαιτεί να κοινοποιούνται τεχνικά εμπόδια στην Κομισιόν. Ε, ε υπάρχει ο οθέτηση νομοθεσία κυρίω κυρίως στον τομέα ε, της επισήμανσης χωρίς κοινοποίηση. Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμόσουν οι αλληλεμποροί αυτές τις απαιτήσει διαφορετικά πληρώνουν βαριά πρόστιμα. Άλλο παράδειγμα λοιπόν ε, μεγάλου προστατευτισμού, αυξημένου προστατευτισμού αυτά ε, δημιουργούν ε, κάποια ωφέλη για τον κατασκευαστή που δραστηριοποιείται ήδη στην εγχώρια αγορά. ας αναφερθούμε τώρα στην ε, νομαθεσία. Με την αναθεώρηση της οδηγίας για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό όλα τα κράτη-μέλη διατηρούν την εθνική προσέγγιση για τη θέση αγαθών σε εμπορία. Έτσι λοιπόν μετακινούν προϊόντα από μία αγορά στη άλλη και οι λαμβάνουν όλη την ευθύνη του παραγωγού για την πληροφορία για τα τρόφιμα. Ο κανονισμό διατηρεί το πεδίο εφαρμογή για αποκλίνουσε εθνικέ ερμηνείε τη ευθύνη του λιανεμπόρου για την πληροφορία των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, ε, συναντήθηκαν ε, δυσκολίες ε, στην Ιταλία για εμπορικούς τρόπους δεν μπορούσε να γίνει επιστροφή του ΦΠΑ άλλο παράδειγμα στην Ισπανία συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής για δύο λοιπάσματα που πολλούνται σε συσκευασία ενός κιλού που δεν απαιτείται σε επίπεδο ευρωπαϊκής αίτησης στην Ιταλία ζητήθηκαν κάποιες δοκιμές για κοινοποίηση εθνικών εργαστηρίων, κάτι που δεν απαιτείται από Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στην Τσεχία υποβάλλεται συγκεκριμένε απαιτήσει για την πώληση αγαθών, όπω ε, παραδείγματο χάρη παιχνίδια για παιδιά κατά των τριών. Δεν υπάρχει σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα μπορούσαμε να συγχυσούμε με τη Γερμανία, όπου το κόστο ε, τη αγορά ε, κρικών συσκευών ε, ήδη περιλαμβάνει το κόστο τη ανακύκλωση. Όταν εξάγονται αυτά τα προϊόντα σε άλλο κράτο μέλο, ε, τότε θα πρέπει να πληρώσει δεύτερη φορά ο λιανέμπορο. Η Γαλλία επιβάλλει η εισαγωγή τυριού να γίνεται σε πακέτο 40 κιλό, ε, ενώ παράγονται πακέτα 15 κιλών. Για να στραφώ στον επιχειρηματικό, στον επιχειρηματικό τομέα έχουμε κάποιες εδαφικές, κάποιους εδαφικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε σε άλλες χώρες ε, ε, προϊόντα με την ίδια τιμή. Η διαφορά μπορεί να έχει αποκλείσει 50% και όταν πρέπει να εξηγήσει γιατί έχουμε τόση διαφορά η εξήγηση είναι «Α, δεν υπάρχει ενιαία αγορά». Και να κλείσω, θέλω να πω, αυτός που χάνει σήμερα από αυτές τις πρακτικές δεν είναι οι ανέμποροι, τελικά είναι οι καταναλωτές. Και γι' αυτό ακριβώ. καλωσορίζουμε το έργο που υλοποιείται σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντουριέ και κάποια από τα ζητήματα τα οποία θίξετε ενδεχομένως να αφορούν και άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα οι πρακτικές σύναψεις συμβάσεων, οι συμβατικές σχέσεις. Δύο άτομα θέλουν να πάρουν αυτή τη στιγμή το λόγο. Δεν ξέρω πόσοι συναδελφοί μου θα ήθελαν να πάρουν το λόγο στο πρώτο τμήμα της Στρογγυλής Τράπεζας. Αρχικά λοιπόν οι επισκέπτες μας, οι προσκεκλημένοι μας και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Ο κύριος Άλφετ Μπουτζάρ από τη Σολντανόσκ θα πάρει το λόγο. Πού βρίσκεστε? Δεν είναι στην αίθουσα, έχει φύγει. Σας βλέπω, ναι, σας βλέπω τώρα. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Εκπροσωπώ την συνδικαλιστική οργάνωση Solidarnosc της Πολωνίας. Η οργάνωσή μου έχει ως μέλη της διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχουμε βέβαια και μία διεθνική συνεργασία. Σήμερα στην Πολωνία υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται από τους εργοδότες. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά στην Πολωνία. Θα ήθελα λοιπόν στην παρέμβασή μου αυτή να επικεντρωθώ στις συνθήκες εργασίας και στα όσα ισχύουν σχετικά με τους μισθούς. Βλέπουμε δυστυχώς ότι οι συνθήκες αυτές είναι δυσχερείς πολλές φορές και οι εργοδότες χρησιμοποιούν μια κλασική δικαιολογία, τον όρο κρίση. Οι εργοδότες λοιπόν επιθυμούν να μειώνουν όλο και περισσότερο το εργασιακό κόστος, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος τώρα να πρέπει να κάνει πάρα πολλές διαφορετικές δουλειές, έχουν αυξηθεί τα καθήκοντά του, ενώ πριν από ένα ή δύο χρόνια τα καθήκοντα αυτά θα γινόντουσαν από ένα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Πώς λοιπόν η κατάσταση αυτή επηρεάζει τους καταναλωτές και πώς επηρεάζει την ε, διεθνή διακίνηση κεφαλαίου. Αναφέρομαι δηλαδή σε διεθνείς παράγοντες όπως οι μεγάλες αλυσίδες ε, σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη επιθυμία εξοικονόμησης χρημάτων. Αυτό όμως έχει αρνητικές επιπτώσεις. Με δύο τρόπους συγκεκριμένα, με δύο σημαντικούς τρόπους. Πρώτον, η ποιότητα των υπηρεσιών που πηγαίνουν προς καταναλωτές. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ε, επιδεινωθεί, έχουν ε, χάσει την αρχική τους ποιότητα. Υπάρχει όλο και λιγότερη ή όλο και φτωχότερη εξυπηρέτηση προς τους καταναλωτές. Στην πράξη, κάθε φορά που ένας καταναλωτής θέλει να καταγγείλει κάτι, έχει παράπονα για ένα προϊόν, για μια υπηρεσία, δεν είναι σε θέση πλέον να απευθυνθεί άμεσα σε μια εταιρεία. Μια άλλη αρνητική επίπτωση είναι ότι οι συνθήκες εργασίας ε, είναι όλο και πιο δυσχερείς. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν εργάζονται για τον ίδιο μισθό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά συνιστούν για μας πολύ σημαντικό πρόβλημα, πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό ενδεχομένως να μην επηρεάζει άμεσα την ροή και την παροχή των ε, αγαθών και των υπηρεσιών, ωστόσο Μιλάμε για μια ενωμένη ενιαία Ευρώπη και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο είναι λογικό οι εργαζόμενοι στο, στην Πολωνία να ζητάνε τις ίδιες συνθήκες εργασίας που έχουν οι εργαζόμενοι σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δύο λεπτά είχατε μόνο στη διάθεσή σας. Η κυρία Βάιλερ θέλει να πάρει το λόγο είναι συνάδελφος από την Επιτροπή μας. Να ζητήσω και τον κύριο Βάντε Βέιντερ από την Εστλέ να μου πει που βρίσκεται στην αίθουσα. Η κυρία Βάιλερ θα πάρει πρώτα το λόγο. Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, να ολοκληρώσετε με σε δύο λεπτά και συνέχεια θα πάρει το λόγο ο κύριος από την Εστλέ. Ε, ναι, πολύ σύντομα. Μία ερώτηση προς έναν από τους ομιλητές μας, τον κύριο Ντουριέ, που είπε ότι σε κάποιους τομείς υπάρχουν ε, ε, εμπόδια από τη μία χώρα προς την άλλη. Ε, κάτι που μοιάζει με ένα στυλ προτεξιονισμού που δεν δικαιολογείται αντικειμενικά όμως. Πριν τρία χρόνια υιοθετήσαμε το λεγόμενο πακέτο αγαθών, το Goods Package και ζητήσαμε τότε αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Όταν ένα κράτος μέλος ε, διατηρεί κάποια μέτρα προστατευτικά που δεν ισχύουν κατά τα άλλα για την αστερική αγορά, θα πρέπει να το αιτιολογεί. Εάν καταφέρει να το αιτιολογήσει επιτυχώς, τότε μπορεί να το διατηρήσει. Το παράδειγμα που ανέφερε ο κύριος Τουριό, κατά τη γνώμη μου, δεν ταιριάζει ε, καθόλου ε, στην περίπτωση αυτή ε, δεν δικαιολογείται αντικειμενικά. Θα πρέπει η Κομισιόν να κάνει κάτι για το θέμα αυτό. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. και ω ασκιώδη ηγητή το είχα πει αυτό και το ξέρω κύριο Ντουριέ. Χρειαζόμαστε περισσότερε εταιρείε οι οποίε θα πρέπει να παραπονεθούν για το ζήτημα αυτό και να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά γιατί έχουν τη νομική ικανότητα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένω όμω ο κύριο Ντουριέ να θέλει να απαντήσει και σε κάτι ακόμα. Είδαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει ήδη οι λιανοπολιτέ επιβάλλουν κάποιου όρου στου προμηθευτέ του οι οποίοι σε πολλέ περιπτώσει δεν τυχαίνουν αμοιβέ αναγνώριση. Δεν υπάρχει αμοιβέ αναγνώριση για κάποια προϊόντα τα οποία φορτώνται σε μια χώρα και διοχετεύονται σε μια άλλη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η αναγνώριση αυτή, η αμοιβέ αναγνώριση και επ' αυτού θα μπορούσε να επιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βέτερ τώρα θα ήθελε να πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι η συγγήτρια έθεσε τα ζητήματα αυτά ως ζητήματα προτεραιότητα στην έκθεσή της για την ε, λιανική αγορά. Η εταιρεία μου ε, ανέκαθεν υποστήριζε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ολοκληρώσει την ε, ενιαία αγορά για τα προϊόντα. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι η αρχική πρωτοβουλία έχει χάσει τον δυναμικό χαρακτήρα που είχε στην αρχή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί για μας πρόβλημα. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, Υπάρχουν ε, αποκλίνουσες ρυθμίσεις ακόμα και εμπόδια όσον αφορά την πιστοποίηση προϊόντων σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Επίσης, ε, σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι κανόνες όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τρίτον, φορολογία όσον αφορά τα τρόφιμα, καθώ επίση και αυθαίρετα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση φορολογία για τα τρόφιμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πάρει να μα απασχολεί από την πρώτη Ιανουαρίου στη Φιλανδία. Τέταρτον, διαφορετικοί κανόνε επιβολή του νόμου. Καθότι υπάρχει μια αποκλίνουσα εναρμόνιση αυτή τη στιγμή τη κοινοτική νομοθεσία, ιδίω όσον αφορά τι ενστάσει τα παράπονα. Τα ζητήματα αυτά καλούμεθα εμεί σε καθημερινή βάση να τα αντιμετωπίσουμε και η εταιρεία μου την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχε στο ανώτατο φόρουμ για την αλυσίδα εφοδιασμού για τα τρόφιμα και αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν μέσω του σχεδίου δράση του δικού σα να καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα αυτά, γιατί οδηγούν σε μειωμένη αποτελεσματικότητα και για τι εταιρείε και για του λενοπολιτέ. Σα ευχαριστώ πολύ για τι αφή σα ε, δηλώσει. Ευχαρίστω να λάβουμε και τα γραπτά σα σχόλια για να τα διανύμουμε και να τα θέσουμε και στην ιστοσελίδα μα. Νομίζω ότι δεν, θέλουν να... δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο στο στάδιο αυτό. Η κυρία Ρουίλε, παρακαλώ. Ε, Πολύ σύντομα. Ε, εγώ αφενός θα ήθελα τον κατάλογο των εμποδίων αυτών στο ε, εμπόριο και να σταλεί ο κατάλογος στην Κομισιόν και όσον αφορά τον κανονισμό περί συσκευασιών Ό,τι προβλήματα δημιουργούνται εδώ είναι προβλήματα και για τους ε, καταναλωτές. Ε, στα κράτη-μέλη βλέπουμε συνέχεια να μην ε, τηρούνται οι κανόνε σχετικά με το μέγεθο τη συσκευασία ώστε να μην ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτή. Θα πρέπει αυτό να, το επισημάνουμε και στον καταναλωτή και στον ε, πολιτή. Ναι. Ωραία. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να καλέσουμε τους κυρίους Χέντριξ και Ντυριά να απαντήσουν στα σχόλια αυτά. Αν μπορείτε παρακαλώ μέσα σε δύο λεπτά θα μας βοηθούσατε. Παρακαλώ κύριε Χέντριξ. Παρακαλώ θέλετε να απαντήσετε και να κάνετε κάποια τελευταία σχόλια. Θα είμαι πολύ σύντομο πρόεδρε γιατί στην πραγματικότητα δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Νομίζω ότι ο κατάλογος των εμποδίων είναι μακροσκελής. Και για το λόγο αυτό δεν έκανα καν απόπειρα να τα αναφέρω στα πέντε λεπτά που είχα. Είναι πολύ πλοκό το θέμα αυτό, πρέπει να το δούμε λεπτομέρως. Το αναφέρω και ο κύριος Διριέ. Λόγου χάρη οι Ιλιανέμποροι υποχρεούνται να αγοράσουν στην ίδια τους τη χώρα και όταν ε, παραδείγματο χάρη βρίσκουν ένα φτηνότερο προϊόν σε άλλη χώρα, δεν επιτρέπεται να το αγοράσουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ προσεκτικά γιατί υπάρχει κάτι τέτοιο, ποιοι είναι οι λόγοι. Από την άλλη για του μικρού λιανοπολιτές ε, αυτό είναι πρόβλημα γιατί οι μικροί λιανέμποροι είναι τμήμα ενό δικτύου συνήθω και επομένω το δίκτυο κάνει όλε τι επαφέ όταν ε, στις μικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται να αγοράσουν ε, μία ποσότητα ίδιες ε, δεν είναι οικονομικά εφικτό ούτε είναι δυνατό για αυτές να αρχίσουν να ψάχνουν σε ένα μπακάλικο παραδείγματος χάρη μπορεί να έχετε πολλά προϊόντα δεν μπορούμε μόνο μένα να ψάχνουν σε όλη την Ευρώπη για το πιο φθηνό προϊόν έτσι λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε αυτό το θέμα της διαφοράς των τιμών αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν μπορούμε να, κάνουμε γενικά να βγάζουμε γενικά συμπεράσματα. Ορισμένε φορέ υπάρχουν ε, καλοί λόγοι για τη ε, διαφορά στι τιμέ, ενώ σε ορισμένε περιπτώσει δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ, κύριο Στυρία. Για τον πρώτο μιλητή από τη Solidar Νόσκ ε, αναφέρετε κι εσείς ότι υπάρχει επικοδομητικός διάλογος στην Ευρώπη και κάτι σημαντικό που τονίσαμε είναι το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματική ενιαία αγορά. Μια άλλη πτυχή που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι η εξή. Εμείς ε, ζητάμε, απαιτούμε να μειωθεί το κενό ε, μεταξύ του κόστος πληρών εταιρεία και του χρήματος που καταλαμβάνει, μάλλον και των χρημάτων που καταλαμβάνει ο υπάλληλος Ρωτήσατε για τις συνέπειες στους καταναλωτές από ε, την κατάσταση που κυριαρχεί στη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο ε, καταναλωτής ε, στην Πολωνία ήταν ε, που είδε ότι μειώθηκε σημαντικά ο πληθωρισμός τα τελευταία 18 χρόνια και η ποιότητα και η η ποικιλία που υπάρχει σήμερα στα τρόφιμα δεν συγκρίνεται με 18 χρόνια πριν και μάλιστα έχουμε αλλαγές στο λιανεμπόριο, ε, δηλαδή σε πολλές ε, περιπτώσεις έχουμε ακόμη και self-service. Ε, όμως είμαι σίγουρος ότι ο ανταγωνισμός θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες και σύντομα. Σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο για τα αγαθά το γνωρίζουμε αυτό και ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και κοινοποίηση. Τώρα, για τον συνάδελφο από την Εστιλέ, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη συνεδρία. Προ... Αυτού όμως θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι έχουμε και μετάδοση στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να καλωσορίσω και όσους μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο, εκατοντάδες ή χιλιάδες μπορεί να είναι. Αν ε, μας παρακολουθείτε ε, μέσω της ε, ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν έχετε καυτά ζητήματα για μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής μας, της Επιτροπής ΙΜΚΟ, και εκεί θα δείτε ποια είναι και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αν μας στείλετε ένα email με μια σύντομη ερώτηση, εγγυώμαι ότι θα φτάσει σε μένα. Έτσι λοιπόν, παρακαλώ να το έχετε κατά νου. Τώρα, για την επόμενη συνεδρία θα έχουμε μια διαφορετική σύνθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε δύο εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι θα αναφερθούν ε, σε θεματικές που είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν να κάνουν ε, με τις εμπορικές και τις συμβατικές πρακτικές τις σχέσεις B2B μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή στο λιανεμπόριο. Έχουμε τον κύριο Ζιλ Στίκ, ο οποίος είναι καθηγητής δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν. Έχει εργαστεί πάρα πολύ στον τομέα αυτό, τον καλωσορίζουμε. Και έχουμε και τον ε, δόκτωρα Πίτερ Ντέβιτ, ο οποίο ε, είναι αναπληρωτή ε, πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όπω πολύ γνωρίζετε, έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία για θέματα για. Ε, που αφορούν την αγοραστική δύναμη και αφορούν ε, τον τομέα των σούπερ μάρκετ και των μπακάλικων. Έτσι λοιπόν, ε, ο καθένας ε, θα έχει 10 λεπτά και νομίζω ότι υπάρχουν διαφάνειε και κατόπιν θα έχουμε και συνεισφορές πέντε λεπτών από τη Μέλα Φρουέν, που είναι Γενική ε, Διευθύντρια ε, του Συνεργασμού για το, το ΕΤΑ και τα τρόφιμα, Αλάν Καλάνσκι, από την Ένωση Εμπορικών Σημάτων και το Πολ Σκέν, ο οποίος ε, είναι Διευθυντής τη Ευρωπαϊκή Τρογγυλής Τράπεζα για το Λιανεμπόριο. Έτσι λοιπόν θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Στίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ζήτημα το οποίο ετέθη σε μένα είναι αρκετά απλό. Μέσα σε 10 λεπτά μπορώ να σας παρουσιάσω το πόρισμα της έρευνάς μου. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν χρειαζόμαστε κοινοτική νομοθεσία για θέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων ή αν αρκεί απλώς νομοθεσία αντιτράστ, δηλαδή το δίκαιο περί Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να δούμε τι υφίσταται σε νομικό επίπεδο, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όλοι γνωρίζουμε, πιστεύω, ή τουλάχιστον το γνωρίζετε εσείς εδώ στην Επιτροπή αυτή, ότι η Οδηγία 29 του 2005 για τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αναφέρεται στα ζητήματα αυτά και εδώ πέρα ο νομοθέτης αναφέρεται στις μεταξύ των επιχειρήσεων αθέμητες πρακτικές και λέει ότι θα μπορούσε να ληφθεί κοινοτική δράση στον τομέα αυτό. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι υπάρχει μία ακόμα οδηγία, μία ανοποιητική οδηγία 114-2006 για τη συγκριτική και την παραπλανητική διαφήμιση μεταξύ επιχειρήσεων πάλι. Και εδώ πέρα ζητάτε ελάχιστη εναρμόνιση όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση και πλήρης εναρμόνιση όσον αφορά την συγκριτική διαφήμιση. Επομένω, ε, έχουμε εδώ πέρα δύο νομοθετήματα για το ζήτημα το οποίο εξετάζουμε. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν διαφορετικέ παραδόσει. Έχουμε τη γερμανική σχολή που ακολουθούν χώρε όπω η Αυστρία και το Βέλγιο, όπου υπάρχει νομοθεσία για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νομοθεσία όμω που δεν υπάρχει σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει, για παράδειγμα, στο αγγλικό δίκαιο, δεν υπάρχει στην αγγλική νομοθεσία. Πρόκειται λοιπόν για εθνικέ πράξεις ανταγωνισμού μεταξύ των ε, επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό παράδειγμα που έχουμε για μια τέτοια νομοθεσία είναι το γερμανικό δίκαιο. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ παλιά νομοθεσία του 1900-1904 ε, που αναφέρεται και στον ανταγωνισμό καθώς επίσης και στα συμφέροντα των καταναλωτών. Και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, εξέλιξη. Η νομοθεσία αυτή εκμοντερνίστηκε το 2004. Αν δούμε τώρα, την, αν κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση στην εναρμόνιση των νομοθετημάτων αυτών, έχουμε καταρχάς ε, την ε, οδηγία 84-450, Έχουμε επίση την οδηγία του 2006 για την παρεπλανητική και συγκριτική διαφήμιση. Και αυτά είναι τα μόνο νομοθετήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια εναρμονισμένη νομοθεσία όσον αφορά τον τον ανταγωνισμό. Το 1965 το Κέντρο Μελετών Max Planck έκανε μία μελέτη για τη δυνατότητα εναρμόνιση τη νομοθεσία για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο και αν είναι δυνατό. Ας εξετάσουμε καταρχάς την ομολογία του δικαστηρίου στα πλαίσια του UCPD. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην υπόθεση C304-08 όπου λέγεται ότι η οδηγία για τις αθέμητες πρακτικές έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής και δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε απλώς σχέση B2B ή μπορούμε να έχουμε και σχέση B2C, δηλαδή επιχείρηση προς καταναλωτή και ισχύει στις περιπτώσεις που αυτό προσβάλλει μόνο τα συμφέροντα του καταναλωτή. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, απαγορεύεται να γίνει μία ανακοίνωση μείωση των τιμών τρει εβδομάδε που ξεκινήσει η περίοδο των εκτόσεων, το καλοκαίρι για παράδειγμα. Ενδεχομένω να πει κανεί ότι αυτό εξυπηρετεί μόνο του ανταγωνιστέ και ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καλείται όμω να εποφανθεί επί του στήματο αυτού και θα μπορέσει να ερμηνεύσει καλύτερα το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για τον αθέμητο ανταγωνισμό όσον αφορά τη διαφήμιση. Επίση υπάρχουν κάποιοι κατά περίπτωση κανόνε στα πλαίσια τη οδηγία UCPD 2. Πάλι εδώ πέρα έχουμε μία υπόθεση που ήρθε στο δικαστήριο από το Βέλγιο για το αν θα μπορούσε να ισχύσει η οδηγία αυτή στην περίπτωση που γίνεται παράλληλη προώθηση προϊόντων. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, διατάξεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί ουσιαστικά από το δικαστήριο και βλέπουμε πολλές φορές ότι οι ανταγωνιστές ουσιαστικά προσφεύγουν κατά τις οδηγίες αυτής κάθε φορά που υπάρχουν περιπτώσεις συγκριτικής ή παραπλανητικής διαφήμισης. Και πάλι λοιπόν τίθεται το ζήτημα αυτό της εφαρμογής της οδηγίας αυτής όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων. Η σχέση τώρα μεταξύ της, το, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που δεν έχει εναρμονιστεί και του, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού όπου υπάρχει μια εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο. Τώρα, ο καονισμός του 2003, υπαριθμών 1, που αναφέρεται στα άρθρα 3 σημείο 2 και 3 σημείο μας λέει σχετικά με τον αθέμητο ανταγωνισμό ότι επί της αρχής δεν μπορεί κανείς στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας να απαγορεύσει αυτά τα οποία επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναλάβουν δράση είτε στα πλαίσια της νομοθεσίας όπως αυτή υφίσταται στη Γερμανία ή στην Γαλλία, αρκεί να μην υπάρχει κριτική μεταχείριση, ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εθνική νομοθεσία που υπάρχει για κατάχρηση δεσπόζουσας θέση. Επίσης λέγεται ότι σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί κανείς να γίνει πιο αυστηρός ή να προχωρήσει σε μέτρα αποκλεισμού σε σχέση με τα όσα ισχύουν σε κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχει επίσης ε, ένα άλλο στοιχείο το οποίο το ξεχνάμε. Στα πλαίσια του αθέμητου ανταγωνισμού εξετάζουμε όλο και περισσότερο νομοθεσία που υπάρχει για ε, τα πνευματικά δικαιώματα. Έχουμε την προστασία των δεδομένων. Έχουμε διάφορα προγράμματα προστασία των δεδομένων στη χρήση που γίνεται στην πληροφορική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πεδίο εξέταση αυτή τη στιγμή διευρύνεται όλο και περισσότερο στην αφορά τι αθέμητε πρακτικέ. Αν δούμε το άρθρο 5, παράγραφος 5 τη Οδηγία 95 του 2008, βλέπουμε ότι στα πλαίσια της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων προβλέπονται κάποιοι νόμοι που έχουν να κάνουν με τις αθέμητε πρακτικές, των αθέμητο ανταγωνισμό. Προχωρούμε λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα ή αναγκαιότητα θέσπιση κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό. Έχουμε πάλι νομολογία του δικαστηρίου για την δυνατότητα ε, θέσπιση μια τέτοια νομοθεσία βάσει της ε, υπόθεσης C380-03 για τα προϊόντα καπνού. Αν είναι να εναρμονιστεί η σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι όντω υπάρχουν εμπόδια στο διακοινωτικό εμπόριο εξαιτία των αθέμητων πρακτικών και του αθέμητου ε, ανταγωνισμού. Διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει βάση προκειμένου να θεσπιστεί κοινοτική νομοθεσία. Επίση, έχουμε και την υπόθεση Cassis de Dijon, όπου λέγεται εδώ πέρα ότι ε, οι εμπορικές πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν σε ορισμένε περιπτώσει βάση για τη θέσπιση νομοθεσία σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να εξαλειφθούν οποιαδήποτε εμπόδια μπορούν να υπάρχουν, να εξαλειφθεί ο του συνταγωνισμού. Αυτά είχα να σα πω. Ο πρόεδρο ε, ζητά να μιλάει ο μιλητή λίγο πιο αργά μετά από αίτημα των διερμηνέων. Φτάνω στα συμπεράσματά μου, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα επαρκές, ε, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να θεσπιστεί κοινοτική νομοθεσία και κυρίως για τέσσερις λόγους. Καταρχάς, το ευρύ πεδίο εφαρμογή της UCPD, όπως το εξήγησα, αφήνει ένα πολύ μικρό περιθώριο για τη θέσπιση ειδική νομοθεσίας για τις εμπορικές πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων. Δεύτερον, οι υφιστάμενοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εμπορικές πρακτικές B2C θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ ανταγωνιστών. Τρίτος λόγος στον οποίο αναφέρθηκα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των, δι... των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τέταρτον, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι η απουσία κανόνων σε ορισμένα κράτη-μέλη και η παρουσία κανόνων σε άλλα κράτη-μέλη ή οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ των κρατών μελών οδηγούν εμπόδια τα οποία οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η πρότασή μου λοιπόν θα ήταν η ακόλουθη να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της UCPD προκειμένου να καλύπτει όλες τι περιπτωσει b B2C και επίσης θα μπορούσαν να προβλεφθούν επιπρόσθετοι κανόνες όσον αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό Θα ήταν δυνατό να θεσπιστούν βέβαια οι ε, κανονισμοί αυτοί, αλλά κατά την άποψή μου δεν θα ήταν ευκταίο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί επιπλέον τέτοιοι κανονισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό του ανταγωνισμού και αυτό στη συνέχεια θα ε, οδηγούσε σε προβλήματα όσον αφορά την υλοποίηση του, ε, της νομοθεσίας αντιτράστ και ενδεχομένως οι κανόνε αυτοί να διέφερναν περισσότερο την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πέρα από την αρμοδιότητα τη κοινωνική νομοθεσία και κάτι τέτοιο δεν θα ήταν επιθυμητό also ε, σας ευχαριστώ που τηρήσατε τα ε, 10 λεπτά και που είχατε μια τόση πλήρη παρουσίαση ε, στα 17 λεπτά. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή. Περιμένουμε πρώτα τις διαφάνειές του. Ε, σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με μία σύντομη εισαγωγή. Ε, μετά, μετά από τις παρατηρήσεις του προηγούμενου ομιλητή, η ε, μελέτη για τα είδη παντοπολίου ήταν μια μελέτη που αποτελούσε μέρος μιας γενικότερης έρευνας ε, που αφορά ένα μέρος του δικαίου περί ανταγωνισμού ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, το φάσμα εδώ είναι ευρύτερο από το φάσμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί Το καθεστώς μας εξετάζει την απόδοση του συνόλου των αγορών και όχι την συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Κατά τον σχεδιασμό λοιπόν ε, διορθωτικών μέτρων εξετάζουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών καθώς και την όλη δομή μιας συγκεκριμένης αγοράς. Νομίζω ότι μπορώ να περάσω κάποιες διαφάνειες και να περάσω στην περίληψη των συμπερασμάτων ε, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν έχω πολύ χρόνο για να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά γενικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού σκοπεύει να εξετα... Ε, ε, εξέτασε μάλλον ε, τις συνθήκες στην αγορά ειδών παντοπολίου και εξέτασε πολλές πτυχές την εξέτασε πολλές πτυχέ ε, και είδαμε ότι τελικά κάνει αρκετά καλή δουλειά η αγορά αυτή όσον αφορά το αποτέλεσμα της ε, προς τον καταναλωτή. Δύο ε, θέματα προέκυψαν. Το ένα ήταν οριζόντιο. Σε κάποιους τομείς υπάρχει πολλή συγκέντρωση στις τοπικές αγορές και εμπόδια για την είσοδο στην αγορά και το δεύτερο θέμα είναι το αποτέλεσμα της ε, δύναμης ε, του αγοραστή. όταν ε, συνδυάζεται με την ανικανότητα να συντάξει κανείς συνθήκες που να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Μια καθυστέρηση, μια παρακράτηση ε, προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα στην ε, αλυσίδα προμήθειας. Ω ε, ως αποτέλεσμα των δύο αυτών θεμάτων που εντοπίσαμε, καταλήξαμε σε κάποια στοχευμένα διορθωτικά μέτρα. Ε, η Επιτροπή μας εξέτασε την ε, λιανική αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο για ε, τα είδη παντοπολίου. Δεν θα πρέπει να γενικευτούν τα συμπεράσματα αυτά για άλλες χώρες, ούτε καν για άλλες αγορές λιανικής εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα από τα μαθήματα της οικονομίας είναι ότι οι λεπτομέρειες έχουν σημασία όσον αφορά την απόδοση των διαφορών αγορών. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Γενικά η ε, άσκηση της ε, δύναμης του αγοραστή οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα. Ε, για παράδειγμα, χαμηλές τιμές, πράγμα θετικό για τον ε, καταναλωτή, μπορεί να οδηγήσει όμως και σε παροχή μικρότερων ποσοτήτων, πράγμα που είναι κακό για τον καταναλωτή. Και η Επιτροπή μας εξέτασε τρεις λόγους γιατί η δύναμη του αγοραστή μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα στην λιανική αγορά. Εγώ εγώ θα αναφερθώ μόνο σε μία από τις τρεις περιπτώσεις ε, που είναι οι αρνητικές επιπτώσεις ε, στα κίνητρα για επενδύσεις εντός ε, του της αλυσίδας προμήθειας. Έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω λίγα από τα στοιχεία που συνέλεξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πλαίσια μιας έρευνας πολυσέλιδης με πολύ αναλυτικές πληροφορίες. Παρακαλώ η επόμενη διαφάνεια. Γενικά, όταν κοιτάμε τη δύναμη του αγοραστή, εξετάζουμε τα στοιχεία από έρευνες. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ότι οι μεγάλοι λιανοπόλητες ε, αγόρασαν τα προϊόντα πιο φθηνά από τους ε, προμηθευτές τους. 100.000 email εξετάσαμε μεταξύ ε, δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ε, και τους προμηθευτές τους, ε, την Άστα και την Τέσκο και το αποτέλεσμα των email αυτών ήταν ότι βρίσκονταν σε πολύ ισχυρή θέση οι μεγάλοι αυτοί λιανοπολιτέ κατά τι διαπραγματεύσει με του προμηθευτέ του. Εξετάσαμε επίση στοιχεία τιμών όγκου και είδαμε ότι Εξετάσαμε τα στοιχεία αυτά σε ένα διάστημα πενταετίας ε, και ε, εξετάσαμε ε, προϊόντα που αντιπροσωπεύουν 1,8 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Περίπου το 2% των συνολικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για είδη παντοπολίου. Εξετάσαμε λοιπόν όπως σας είπα μια σειρά πιθανών μέτρων ε, όσον αφορά την, τον καθορισμό των τιμών ε, και ποια ήταν τα συμπεράσματά μας. Τα βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, είδαμε την μέση τιμή που πληρώνεται από τους τέσσερις μεγάλους λιανοπολιτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τους προμηθευτές τους στη διάρκεια του χρόνου. Βλέπετε την κάτω γραμμή στο διάγραμμα αυτό ε, και στα, ε, ανα πάσα στιγμή στα πέντε αυτά χρόνια οι τέσσερις μεγάλοι ε, λιανοπολιτές πληρώνουν χαμηλότερες τιμές προς τους προμηθευτές τους από ότι άλλοι λιανοπολιτές, μικροί χοντρέμποροι και οι άλλες ενώσεις. Από τις διάφορες κατηγορίες των συμμετεχόντων βλέπετε τις ομάδες που πληρώνουν χαμηλές τιμές, άλλες κατηγορίες ε, παραγωγών όμως ε, πληρώνουν και κατά καιρού χαμηλές τιμές. Το μάθημα που μάθαμε από αυτό είναι ότι η δύναμη του αγοραστή δεν ε, συνδέεται αποκλειστικά με το μέγεθος του ελιανοπολιτή. Έχει να κάνει και με την δυνατότητα διαπραγμάτευσης χαμηλών τιμών από τους προμηθευτές τους. Μικροί λιανοπόλητες ε, κατά καιρούς μπορούν να ε, ε, αλλάξουν προμηθευτές πιο εύκολα και έτσι μπορούν να πετύχουν χαμηλότερες τιμές. Το τρίτο συμπέρασμα από την ανάλυση αυτή ήταν ότι το αποτέλεσμα της κλίμακας όσον αφορά τις τιμές το αποτέλεσμα ήταν ε, πολύ μικρότερο όσον αφορά γνωστές μάρκες. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένη εταιρεία, ε, σκεφτείτε όμως ένα προϊόν σαν την Coca-Cola ή την Pepsi-Cola. Τρία μαθήματα λοιπόν. Οι μεγάλοι λιανοπολιτέ πληρώνουν λιγότερα. Το μέγεθο του λιανοπολιτή ε, δεν είναι ο μόνο παράγοντα που ορίζει την δύναμη του αγοραστή και ε, τρίτον, οι τιμές που διαμορφώνονται έχουν πολύ λιγότερη σχέση με το μέγεθος του λιανοπόλητη εάν τα προϊόντα αυτά είναι γνωστής μάρκας. Η δύναμη του αγοραστή φαίνεται Σαφώ ε, καθώ και κάποιες από τις δυνάμεις που οδηγούν στη δύναμη του αγοραστή. Ωστόσο, η δύναμη του αγοραστή από μόνη ε, δεν ε, οδηγεί αυτομάτως σε... το, το ότι οδηγεί η, αγοραστική δύναμη, η δύναμη του αγοραστή σε χαμηλότερες τιμές, αυτό γενικά είναι καλό, όχι πάντα όμως. Ο λόγος που κάποιες τέτοιε χαμηλέ τιμέ μπορεί να είναι επιζήμιε για τον καταναλωτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέτασε κάποιους τρόπους που μπορούμε να έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή. Ε, είδαμε ε, το, τον συνδυασμό της ε, μη πληρότητας των συμβάσεων και την εκ των υστέρων καθυστέρηση ή μη τήρηση της σύμβασης. βλέπετε εδώ την επόμενη διαφάνεια. Πολλέ από τι περιπτώσει αυτές έχουν να κάνουν με αναπάντεχο κόστος ε, ή με υπερβολικούς κινδύνους. Ε, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ε, ο υπερβολικός κίνδυνος μπορεί να έχει να κάνει με τον κίνδυνο κλοπής από την αποθήκη, θέματα ασφάλειας της αποθήκης του Λιανοπόλητη. Εξετάσαμε το θέμα των αναδρομικών πληρωμών είναι στοιχεία που φαίνονται και σε άλλε ε, έρευνες, ε, όπως για παράδειγμα μια έρευνα που θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου, μάλλον θα πρέπει να ε, πάω κατευθείαν στα συμπεράσματά μου. Στα πλαίσια της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού είδαμε σαφώς να, υπάρχει, να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την δύναμη του αγοραστή. Υπήρχαν Αποδείξει ότι μια σύμβαση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Ε, είδαμε και το θέμα της ε, αναδρομικής προσαρμογής ε, των τιμών. Υπάρχουν δηλαδή κάποια αναπάντεχα γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την δυνατότητα των προμηθευτών να παρέχουν τα προϊόντα. Ε, ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού ε, εισήγακε και έναν κώδικα ε, δεοντολογίας, έναν κώδικα πρακτικής ε, και προτείναμε και στην κυβέρνηση να ε, δημιουργήσει μια θέση διαμεσολαβητή για να λύνονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στα πλαίσια του κώδικα αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα σας ε, επέτρεπα να συνεχίσετε, διότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μα είπατε. Κυρίες και κύριοι, όμως έχετε ε, αντίγραφο των διαφανειών αυτών. Μπορείτε λοιπόν να τα εξετάσετε. σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντέιβι. Uh, λοιπόν, να προχωρήσουμε. να ακούσουμε κάποια πεντάλεπτα σχόλια. Θα καλέσω την κυρία Φράουεν, που είναι Γενική Διευθύντρια της Συνομοσπονδίας των Βιομηχανιών ε, Ποτών και Τροφίμων. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία ποτών και τροφίμων της Ευρωπαϊκής είναι πολύ σημαντικό που είμαστε εδώ το θέμα των συμβατικών και εμπορικών πρακτικών στι σχέσει μεταξύ επιχειρήσεων. Είναι ένα θέμα που έχει προκύψει στην αλυσίδα τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Όλοι ξέρουμε γιατί. Όλα ένα και μεγαλύτερη εστίαση δόθηκε στι σχέσει ε, μεταξύ τη αλυσίδα, κατά μήκο τη αλυσίδα, κυρίω με την ε, με το λιανεμπόριο από τη στιγμή που συστήθηκε η ομάδα υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα του τομέα το και τροφίμων στην Ευρώπη. Υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις σε αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ορθή λειτουργία της διατροφικής αλυσίδα. Αυξήθηκε το ενδιαφέρον, έχουμε ένα νέο φόρουμ υψηλού επίπεδου και δημιουργήθηκε μια ειδική πλατφόρμα αφιερωμένη σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, καθώ υπάρχει τόσο ενδιαφέρον, φαίνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. επίση ο Επίτροπο Μπαρνιέ ανέφερε τι θέματα συμπορικέ πρακτικέ σε πολλέ πρόσφατε ομιλίε του και ανέφερε την ανάγκη να βελτιωθούν σχέσει κατά μήκο τη αλυσίδα και εσείς κυρία Κορέτσα Μπίλτ, το Single Market Act που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2010. Εδώ η Κομισιόν αναφέρει την ανάγκη για δράση κυρίως στον τομέα ε, των τροφίμων η ΕΟΚΕ αναφερθήκε σε αυτό το θέμα. Ε, υπήρξαν και πολλέ άλλε δηλώσει, μελέτε κτλ. Και όλα αυτά υπογραμμίζουν ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, έχοντα αυτά κατά νου και επειδή μας ε, ζητήθηκε από διάφορες γαμαδέλτα της Κομισιόν ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα για το τι πράγμα μιλάμε. Εμείς αποφασίσαμε να εξετάσουμε στενότερα το ζήτημα αυτό και αποφασίσαμε να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για να μάθουμε περισσότερο τι συμβαίνει. Έτσι, βάσει των βέλτιστων πρακτικές ε, αναπτύξαμε ε, ένα μικρό κατάλογο για αθέμητες πρακτικές. Ε, πρόκειται για ένα πάγιο κατάλογο, αλλά εμεί θέλαμε να δούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αν είναι βρεώστε δεδομένο, αν περιορίζεται σε κάποια κράτη-μέλη, αν είναι εξαιρετικές αυτές τις περιπτώσεις ή αν προκύπτουν συχνά, ποιο είναι το μέγεθος των εταιριών που θίγονται κτλ. Έτσι, έτσι, έτσι λοιπόν ε, ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη και κάλυψε πάνω από τα μισά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμμετείχαν σε αυτά αρκετά μεγάλα αλλά και μικρά κράτη-μέλη και κάποια κράτη-μέλη όπου είχαμε η νομοθεσία ή όπου υπάρχει ε, ένας εθελούσιος κώδικας. Ήδη έχουμε λάβει πάνω από 600 απαντήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο που στείλαμε μόλις το Δεκέμβριο. Και νομίζω ότι αυτό δηλώνει ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Οι απαντήσεις προήρθαν και από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν φυσικά ότι υπάρχει πρόβλημα. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσει που έστειλαν τι απαντήσει του είπαν ότι είναι εκτεθειμένε ε, σε έξι είδη ε, αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Ε, Εμεί είχαμε ένα κατάλογο 12 και είπαν, αυτές αναφερθήκαν σε 6 κατά το 2009. Βέβαια στις απαντήσεις ε, δεν κατονομάζουν ε, κάποιους λιανοπολιτές, ε, δεν θέλουμε να δακτυλοδεικνύουμε κάποιους. Δυστυχά σήμερα δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εργασία μας, δεν είχαμε το χρόνο να προβούμε σε πλήρη ανάλυση και θέλουμε να έχουμε προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Όμως θα σας πούμε περισσότερο όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα θα το πράξουμε εγκαίρως για τη συνεδρίαση της πλατφόρμας του Μαρτίου που θα αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στο φόρουμ υψηλού επίπεδου και ευχαριστώ σας παρουσιάσουμε τότε τα αποτελέσματα. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες εταιρείε ε, που απάντησαν μας είπαν ότι ε, δεν ε, είχαν διαμαρτυρηθεί επειδή φοβούνταν ότι μπορεί να υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις ε, και ε, ο λόγος που οι μονομένες εταιρείε τροφίμων φοβούνται να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό και να μιλήσουν είναι ε, γιατί προτίμησα να, να χρησιμοποιήσουν τη δική μου οργάνωση ως εκπρόσωπο Καμία από τις μεμονωμένες εταιρείε δεν συμμετείχε απευθείας στην πλατφόρμα B2B. Δεν συμμετέχουν απευθείας γιατί δεν θέλουν να παρουσιάζεται ότι διαμαρτύρονται έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με επικοδομητικό τρόπο. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι διαφορέ μα, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιε λύσει τι οποίε θα έχουμε συμφωνήσει από κοινού, γιατί και εμεί από κοινού αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα με του λιανέμπορου. Ελπίζουμε ότι η πλατφόρμα αλλά και το φόρουμ θα μα βοηθήσουν να ξεβρούμε λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λύσει αποτελεσματικέ που να μπορούν να εφαρμοστούν και φυσικά και η δική σα άποψη θα μα βοηθήσει βοηθήσει να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, um, ε, εμείς συμφωνούμε με τη συνεισφορά σα. Ευχαριστώ ε, να συνεισφέρουμε, αλλά όπως είπατε είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα και θέτει και προκλήσεις. Ας το θέσουμε έτσι. Ε, Τώρα θα δώσουμε και το λόγο σε κάποιον συναδέλφο που θα έχει, δύο θα, θα έχει την ευκαιρία να μας πει δύο λόγια σχετικά με το γράφο εργασία, Η Άννα Μαρία τοποθετήθηκε πριν σε αυτό. Προηγουμένω ε, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ε, ε, ισχύ που έχουν τα εμπορικά σήματα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Άλαν Γκαλάνσκι, ο οποίος προέρχεται από την Ένωση Εμπορικών Σημάτων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την ε, κυρία Κοράτσα Μπίλ που μας κάλεσε σε αυτή την ε, σημαντική συζήτηση. Δύο λόγια. Ε, να σας πω ότι εμείς εκπροσωπούμε μια μεγάλη γκάμα εμπορικών σημάτων από τη Γερμανία, την Ιταλία, τις σκανδιναβικές χώρες και οι περισσότερες εταιρείες αυτές δεν είναι πολύ μεγάλες εταιρείε, πολλές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι λοιπόν έχουμε μια ποικιλόμορφη εικόνα. Τα επόμενα λεπτά και βλέπω ότι δεν περνάει η ώρα. Πρέπει να βάλετε μπρο και το ρολόι, το χρονόμετρο. Κοιτάξτε, εγώ ούτε ή έχω συνηθίσει να βλέπω το ρολόι γιατί παρακολουθώ μπάσκετ. Έτσι λοιπόν θα παρουσιάσουμε ένα είδος αθέμη της πρακτικής ε, σε λίγο που θίγει την καινοτομία, τα εμπορικά σήματα και την επιλογή των καταναλωτών αν ε, πολύ ψωνίζετε, που είμαι σίγουρος ότι πολύ ψωνίζετε, θα ξέρετε ότι στα περισσότερα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, ε, όταν ε, έχουμε προϊόντα με εμπορικό σήμα, τότε ξέρετε ότι αυτά ανταγωνίζονται και οι λιανέμποροι είναι ανταγωνιστές των κατασκευαστών εμπορικών σημάτων. Όμως, να σας πω ότι οι κατασκευαστές εμπορικών σημάτων δεν έχουν ε, πρόβλημα με το ζήτημα του ανταγωνισμού. Ε, γιατί ο ανταγωνισμός, ε, αν είναι θεμητός, είναι καλός για όλους. Δηλαδή, οι κατασκευαστές συνήθω ζητούν από ένα παραγωγό να βασίζεται στον ίδιο, στον κύριο ανταγωνιστή να πουλήσει τα προϊόντα τους. Και αν θα γίνει κάτι τέτοιο, τι αναμένεται να γίνει στην πράξη. Αυτό μάλλον αναμένεται να γίνει, αλλά συνήθω στην πράξη πολλέ φορέ ζητείται από του κατασκευαστέ να μοιραστούν απόρριτε πληροφορίε με του ε, λιανεμπορού όταν, παραδείγματο χάρη, έχουμε πρόθεση προϊόντων. Ε, Αυτό ο διτό ρόλο του λιανεμπορού ω ανταγωνιστή αλλά και ω πελάτη σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ευθύνη για να διασφαλίσει ότι είναι θεμητό ανταγωνισμό. Από τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης που ανέφερε η ΜΕΛΑ προκύπτει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει πάντοτε αυτό ότι κάποιοι από τους ε, κατόχους εμπορικών σημάτων μας είπαν ότι έχουν δει λιανεμπόρους να χρησιμοποιούν πληροφορίες που απέκτησαν ως καταναλωτής για να αναπτύξουν τη δική τους ανταγωνιστικό εμπορικό σήμα, τη δική τους ανταγωνιστική μάρκα και χρησιμοποίησαν το καθεστώ τους ε, ως πελάτη με έναν τρόπο που δεν είναι διαθέσιμο σε άλλες ανταγωνιστές. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε ίσους όρους, δεν έχουμε level playing field. Και για να χρησιμοποιήσω μια αναλογία από το ποδόσφαιρο, δεν έχουμε τον κατασκευαστή των περικοστινών που ε, παίζει μόνο, ε, αλλά εκτό έδρα, αλλά ε, έχουμε παραδείγματο χάρη και το Ιανέμπορο, σαν να παίζει πάντοτε εντό έδρα και ξέρει από πού θα του έρθει τον γκολ. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι εδώ πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει και διαιτητής. έτσι. Και εδώ η απάντηση του ε, ανταγωνιστή ε, μπορεί να ακυρώσει το πλεονέκτημα που θα έχει ε, ο κάτοχος του εμπορικού σήματος και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους καταναλωτές γιατί έχει επίπτωση στην επιλογή, αλλιώνει την επιλογή. Όμως η πρακτική αυτή δεν είναι καθολική στον τομέα μας και πολλοί ανέμποροι είναι πολύ επιτυχείς στην αγορά χωρίς ε, να ε, παραβαίνουν το απόρριτο. Ε, όμως, πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Και να σας πω τι κάναμε. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι οι λιανέμποροι οι οποίοι ε, κάνουν καλά τη δουλειά του και με του οποίου έχουμε πολύ καλέ ε, σχέσεις συνεργασίας οι ίδιοι θα συμφωνούσαν με το ότι οι, οι πρακτικές στις οποίες αναφερόμαστε είναι καλέ πρακτικέ και πρέπει να ξέρουμε το κίνδυνο αντιτράστ ε, που έχει να κάνει με τι οριζόντιε κατευθυντήριε γραμμέ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω πώς ε, αντιμετωπίζουν αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων οι εταιρείε τι είδου καλές πρακτικές εφαρμόζουν σήμερα σε εκούσια βάση για να αποφύγουν ε, αθέμητη και μη ανταγωνιστική συμπεριφορά ε, με το στόχο να, υπάρχει, να υπάρχουν αναλογικά μέτρα ε, που να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστούν τέτοιες πρακτικές. Οι αθέμητες πρακτικές ε, θίγουν την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας προμήθειας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε αποτελεσματικές λύσεις εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερομένους. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά, προκειμένου να ωφελήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις και τους λιανεμπόρους που ήδη ε, έχουν μια ορθή συμπεριφορά και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και το συμφέρον των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Αλά. Ήσασταν πολύ σαφείς και ε, σεβαστήκατε επίσης και το χρόνο που σας δόθηκε, μόνο ότι είχατε λίγο περισσότερο χρόνο στην αρχή. Προτού ξεκινήσει η γενική συζήτηση, πρέπει να σας πω ότι έχω ήδη τρεις ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή να μου πούν αν θέλουν να πάρουν το λόγο και ποιοι είναι αυτοί. Ο τελικός μας ομιλητής πρώτο ξεκινήσει συζήτηση είναι ο Πολ Σκέαν από, τον, από την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για την Ελληνική Πώληση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Κοράτσα Μπίλ, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή και με τους συναδέλφους μας αλλά και με τους ευρωβουλευτές από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι η MCA ήδη έχει ξεκινήσει μια έρευνα προκειμένου να εντοπίσει τα στοιχεία αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Θεωρώ ότι ε, είχαμε πάρα πολλέ συζητήσεις, κάποια θεωρητικά συμπεράσματα, τα οποία δεν βασίζονταν σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, σε αποδεικτικά στοιχεία. Αρχίζουμε και συλλέγουμε πλέον τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σαφώς υπάρχουν κάποια ζητήματα, το είδαμε αυτό και από αυτά τα οποία είπε η Μέλα και ο Αλά. Πρέπει να σας πω ότι ο τομέας κλινικής πώλησης ε, αντιμετωπίζει προβλήματα και με τον τομέα των προμηθευτών. Βλέπουμε πολλές φορές ότι οι πρακτικές που ακολουθούν η μεγάλη παραγωγή, η μεγάλη διανομή προς τους λιανοπολιτές δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε παραδόσεις οι οποίες είναι μερικές, οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες, που οδηγούν πολλές φορές σε πολύ δυσμενή αρνητικά αποτελέσματα για τον λιανοπολιτή, ο οποίος καλείται να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Επίσης έχουμε έναν κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς, αναφερθήκαμε σε αυτό πριν από λίγο, και έχουμε και ορισμένες μη δικαιολογημένες καθυστερήσεις, ή πολλές φορές πρέπει να επιληθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τιμολόγια και οδηγούν πολλές φορές σε καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τους 12 μήνες. Και βέβαια το χρέος, το κόστος καλείται να καλύψει ο λιανοπολιτής. Συμφωνώ με τη Μέλα και τον Αλάου ότι πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα να επιληθούν και πρέπει αυτό να γίνει με έναν τρόπο θετικό, επικοδομητικό, λογικό. Η Αστρογγυλή Τράπεζα για τη Λιανική Πώληση αποτελεί τμήμα της πλατφόρμας που έχει συσταθεί για τη μελέτη των ε, πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων. Θέλουμε στα πλαίσια της πλατφόρμας αυτής να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε μείωση του ανταγωνισμού και που δεν θα οδηγήσουν σε μείωση της προσφοράς προς τον καταναλωτή. Και νομίζω ότι κάποιε συζητήσει που κάναμε για την αλυσίδα του εφοδιασμού πολλέ φορέ αφήσανε εκτό, παραμέρισαν εντελώ τα συμφέροντα του καταναλωτή. Επίση, χρειαζόμαστε ανεξάρτητα επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα καταφέρουν να ενισχύσουν την ανάλυση την οποία κάνουμε. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο 2009 υπέβαλε μια πολύ λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται σε όλα αυτά τα προβλήματα. Σε τρία σημεία θα ήθελα να αφαιρθώ. Αγοραστική δύναμη. Συμφωνώ μετά όσο είπε ο κύριος Ντέιβις για τη διασύνδεση, την απουσία διασύνδεσης που ενδεχομένω να υπάρχει μεταξύ της αγοραστικής δύναμης καθώς επίσης και του όγκου των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Πάρα πολλέ έρευνε αναφέρονται στην ενοποίηση, την ολοκλήρωση του ε, τομέα λιανικού εμπορίου και βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές η απουσία ενοποίησης, απουσία ολοκλήρωσης του τομέα αυτού έχει να κάνει με τις αθέμετες πρακτικές που υπάρχουν πάρα πολλές ή και με την δεσπόζουσα θέση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και αντικείμενο κατάχρησης. Τώρα, η κλίμακα αυτή καθ' αυτή και αυτό επηρεάζει αν θέλετε τα πράγματα η κλίμακα, η διαφοροποίηση στη μέση είναι κάτι το λογικό. Δεν μπορώ εγώ ω ιδιώτη να αγοράσω μια καρέκλα, για παράδειγμα, στην ίδια τιμή με την οποία θα την αγοράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παραγγέλνει 700 καρέκλε, το μία. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πολύ σημαντική αγοραστική δύναμη. Ο Αλά και η κυρία Κοράτσα Μπίλ στην αρχή αναφέρθηκαν στο εμπορικό σήμα Θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι έχουμε προϊόντα τα οποία φέρουν εμπορικό σήμα. Σαφώ μπορούν να οδηγούν σε κάποιε δυσκολίε. Πάντω είναι προϊόντα τα οποία προστατεύονται από την νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα και διέπονται ουσιαστικά από κανόνες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τον καθορισμό των τιμών και για την πληροφόρηση του καταναλωτή. όσον αφορά το copy-cutting, την ε, αντιγραφή. Νομίζω ότι και εδώ πέρα θα πρέπει να μας απασχολήσουν σε αυτές οι περιπτώσεις παραχάραξης, παραποίησης, απομίμησης που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πολύ συχνά μιλάμε για πραγματική κλοπή πνευματικού δικαιώματος. Δεν θα πρέπει όμως ε, το ζήτημα του copycat να, της αντιγραφής να συγχαίεται με την παραποίηση. Πολλές φορές η αντιγραφή μπορεί να υφίσταται στα πλαίσια της παραγωγής ενός προϊόντος. Είμαστε αθεσί για να συζητήσουμε πιθανές λύσεις, αρκεί όμως να βασιζόμαστε σε απτά δεδομένα, τα οποία θα έχουν συλλεχθεί μέσω ανεξάρτητων ερευνών και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση βέβαια να βαίνουν όλα αυτά κατά των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που ακούμε και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων ε, είναι σειρά σα ε, τώρα να μας κάνετε τι δικές σας παρατηρήσεις. Η κυρία Στάιλερ ζήτησε το λόγο. Θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα ή θέλετε να ακούσουμε πρώτα τους ε, ομιλητές μας από το ακροατήριο. Ωραία, μετά διαβάζω τον κατάλογο των ομιλητών. Πού βρίσκεστε? ο κύριος Μιχαήλ ε, Σπενγκάρο από την ε, Ιταλική Ένωση Παραγωγών Κρέατος είναι παρόν. Ωραία. Και ο κύριος Φάμπιαν Βέινερτ από μια ένωση της Γερμανίας. Υπάρχει άλλος? Μια ερώτηση από το πίσω μέρος της αίθουσας. θα σας δώσουμε ένα έντυπο να σφυλιρώσετε για να γνωρίζουμε ποιος είστε. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τους ίδιου κανόνες με όλους άλλους. Ο κύριος Λάκη λοιπόν πρώτος, ο κύριος Σπαγκάρο και ο κύριος Βέινερτς. Και ο κύριος Μπουτζάρο ζήτησε το λόγο, αλλά ήδη πήρατε το λόγο στον πρώτο γύρο θέλετε, ζητήσατε το λόγο και στον, και στον τρίτο γύρο. Δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο σε, σε κάθε γύρο. Ε, θα δούμε αν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά μου δίνετε για να μιλήσω όχι μόνο για τον τομέα των ε, τροφίμων και των ε, ποτών, αλλά και για τον εναλλακτικό τομέα. 380.000 ε, εταιρείες στην Ευρώπη κατασκευαστές αυτοκινήτων εκπροσωπούμε. Ήμασταν παρόντες και στο φόρουμ σας και στην συνάντηση του Οκτωβρίου και βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με την Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες. Ε, μας ενδιαφέρει ο ρόλος του διανομέα στην ε, Ευρώπη. Δεν εκπροσωπούμε τους κατασκευαστές αλλά τους επισκευαστές και είναι σημαντικό να έχουμε προστασία του καθεστώτος των ε, μελών μας. Γιατί είναι αυτό τόσο σημαντικό, διότι Μέχρι τώρα, μέχρι το 2013 είχαμε έναν κανονισμό που προέβλεπε γενική ε, παρέκκληση, ο οποίος μας παρήχε κάποια ε, προστασία. Ε, ως αδύναμο μέρος στις συμβάσεις που συνάπτουμε με τους κατασκευαστές. Υπάρχει το θέμα των ρητρών ε, στις συμβάσεις μεταξύ κατασκευαστών ε, και ε, εκπροσώπων και κυρία Μπίλτα έχουμε ζητήσει συνάντηση μαζί σας και με τους σκιώδεις εισηγητές και φυσικά και με τον κύριο Χάρμπορ. Έχουμε, συναντούμε κάποια σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τον καθορισμό του, ε, του στόχου πωλήσεων. Ε, εάν δεν πετύχουμε μέχρι το 2013 κάποια άλλη ρύθμιση, θα συνεχίσουμε να είμαστε το αδύναμο μέρος της, της ε, ελπίζουμε ότι πετύχουμε κάποιο επίπεδο προστασία. Σα ευχαριστώ και σα ευχαριστώ που ακούσατε όλοι μα την επιχειρηματολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καθότι είναι ένα τομέα για τον οποίο γνωρίζω πολύ λίγα, θα μιλήσω με την κυρία Κόρα Τσαπίλ σχετικά, ο κύριο Παγκάρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ γρήγορα σε σχέση με το private label, με την ιδιωτική ετικέτα. Γενικού χαρακτήρα σχόλιο. Ό,τι αφορά την ιδιωτική ετικέτα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εκπροσωπώ μια τελική ένωση της Κάνελουκ σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ετικέτα. Προσωπογράφουμε 100% όσοι υπόθηκαν ε, από τον κύριο από τον κύριο Λεγκαλάσκη και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Για την ιδιωτική ετικέτα έχουν πολλά γραφή και υποθεί. Σίγουρα ιδιωτικέ ετικέτες είναι μια πραγματικότητα της αγοράς. Ε, σίγουρα ε, έχουν πάρα πολλές θετικές ε, πτυχές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπογραμμίσω ότι όλα όσο έχουν γραφεί σε σχέση με την ιδιωτική ετικέτα τα τελευταία χρόνια και η πιο σημαντική δουλειά είναι το βιβλίο του Oxford University Press του 2009. Όλα έχουν γραφεί υπογραμμίζουν ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλέ ε, θετικέ πτυχέ του private label, τη ιδιωτική ετικέτα, αλλά τονίζεται επίση ε, ότι εμφανίζονται και πάρα πολύ αρνητικέ πτυχέ που κατά την άποψή μας, αν δεν διορθωθούν εγκαίρως, θα έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Ο κύριος Γκελάσκη ήδη υπενθύμησε κάποια τέτοια θέματα. Εγώ απλώς θέλω να προσθέσω μια ακόμη πτυχή που ξεχνάμε ενίοτε. Το θέμα της μη ορθής πληροφόρησης του καταναλωτή. Γιατί πάντοτε, όλο ένα και περισσότερο, μέσω της ιδιωτική ετικέτας ε, βλέπουμε ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ κάνουν τον καταναλωτή να πιστεύει ότι αυτά είναι που εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, ενώ κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάνουν τον καταναλωτή να πιστεύει ότι αυτοί παράγουν το αγαθό. Αυτό οδηγεί φυσικά ε, στον παραγωνισμό των παραγωγών. Γιατί αν δεν με γνωρίζει ο καταναλωτή, δεν μπορεί να με ε, ελέγξει, δεν μπορεί να, επιλέξει τη δική μου μάρκα και είμαι πιο ευάλωτο έναντι μια σειρά εμπορικών πρακτικών στι οποίε αναφερθήκαμε προηγουμένω. Και μιλώ για θέμητε πρακτικέ. Εδώ θα σταματήσω για την ιδιωτική ετικέτα και ένα γενικό σχόλιο. Έχουμε μιλήσει πολύ για την ε, νέα εξεύρυνση ισορροπίας της αγοραστικής δύναμης στην αγορά. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση για τέτοια ισορρόπηση. Δεν θέλουμε οι συμβατικές ε, ε, εξουσίες να επανισορροπηθούν εμείς. Τι ζητάμε αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής που συμμετέχει και στο φόρουμ. Όμως εμείς τη ζητάμε ίσους κανόνες για όλους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα χρήσιμα σημεία που μας επισημαίνετε και ήμουν γενναιόδωρος, αλλά δεν θα είμαι τόσο γενναιόδωρος για τους επόμενους. Ε, κύριε Βέινετ, παρακαλώ. Two minutes. Yeah. Έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπούμε 400 μέλη από διαφορετικούς τομείς, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα θέλαμε σαφώς και εμείς να έχουμε μια εσωτερική αγορά με ισότιμους θεμητούς κανόνες συνταγωνισμού. Ο κύριος Αλάν Γκαλάσκι αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ζήτημα αυτό. Επίσης, Όταν έρθουμε στην ημερήσια διάταξη στο ζήτημα των επιλεκτικών συστημάτων, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Εδώ πέρα βλέπουμε την προσέγγιση αυτή με μια αρνητική σκοπιά. Ενώ βλέπουμε ότι στη Γερμανία το ζήτημα αυτό έχει λειτουργήσει θετικά. Ας είμαστε λίγο πιο θετικοί, ιδίω έχει οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους παράγοντες στον τομέα της λιανικής πώλησης. Όσον αφορά την ε, ε, όσον αφορά το ευρύ φάσμα των προϊόντων, αλλά και όσον αφορά τον ανταγωνισμό για την καλύτερη προσφορά. Αν εξετάσουμε ιδιαίτερα τον τομέα των καλλιντικών στην ε, Γερμανία, ακόμα και σε κρατήδια με όχι τόσο καλή δομή Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες καλές προσφορές που μπορεί να πετύχει κανείς. Ε, έτοιμά μου λοιπόν προς την εισηγήτρια και όσους ε, συμβάλλουν στον στην έκθεση αυτή είναι να ε, εξετάσουν, να αξιολογήσουν τα διάφορα αυτά συστήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσει που ακούσαμε. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Κοράτσα Μπίλτ τις έχει σημειώσει. Προχωρώ στην κυρία Στάιλερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ήθελα να ρωτήσω τους ε, ομιλητές ε, που μίλησαν για τον ε, τομέα των παντοπολίων τι πιστεύουν σχετικά με την είδηση που ακούσαμε σήμερα ότι ε, οι τιμές των καλλιεργιών θα αυξηθούν ε, από 50 έως 100% τα επόμενα χρόνια. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον τομέα των ε, παντοπολίων. Και επίσης όσον αφορά την αυτορύθμιση και τα προαιρετικά μέτρα λειτουργούν αυτά στην πράξη και τέλος όσον αφορά τις μάρκες πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Πότε μια μάρκα δεν είναι μάρκα όταν ο λιανοπολτής χρησιμοποιεί το δικό του όνομα ως μάρκα και πότε... Μιλάμε για ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων μαρκών, έτσι δεν είναι. Ε, και όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών και όσον αφορά τα μερίδια στην αγορά. Ακούσαμε παρατηρήσεις ε, σχετικά με την αξία των ε, μαρκών. Κάποιοι άνθρωποι θα πληρώσουν παραπάνω για να πάρουν συγκεκριμένη μάρκα, ε, αλλά περνάμε δύσκολους καιρούς. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να, να διστάσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και όπως ξέρουμε στο τομέα της λιανοπολικής η τιμή παίζει σημαντικό ρόλο. Πώς επηρεάζονται λοιπόν οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινεί μεταξύ μας. Ε, επενδύονται χρήματα στις διάφορες ε, μάρκες. Ε, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων μακών θα πρέπει να είναι κάτι θετικό για τους καταναλωτές. Αυτά ήθελα να ρωτήσω και τήρησα και το χρόνο μου βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαχάρο, έχουμε χρόνο εάν περιοριστείτε στο δίλεπτο. Υπάρχει άλλος που ζητάει το λόγο. Αν θέλετε να περιοριστείτε σε, στα δύο λεπτά, σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο ζήτημα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Μέχρι στιγμή δεν υπόθηκαν σπουδαία πράγματα για το ζήτημα αυτό, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα λεπτό και ευαίσθητο. Κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πετυχαίνουν πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα χάρη στους πολύ χαμηλούς μισθούς που πληρώνουν και βρίσκονται επομένως σε πολύ ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Για παράδειγμα, στην Πολωνία ένας ταμείας κερδίζει 300-400 ευρώ το μήνα. Μικτά μάλιστα. Ξέρετε ποιοι είναι οι μισθοί βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, δεν άγει να σα το πω αυτό. Συχνά λοιπόν οι εργαζόμενοι αυτοί λειτουργούν στα πλαίσια πολύ αρνητικών συμβάσεων, καθόλου ευνοϊκών για τους ίδιους. Είναι συνήθως συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θεωρώ ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι συνθήκες εργασίας αποτελούν κοινωνικό τάμπινγκ, θα πρέπει να εξαλειφθούν αυτές οι συνθήκες εργασίας και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό εργαζόμενοι για καλύτερες και πιο ποιοτικέ θέσεις εργασίας, για καλύτερους όρους εργασίας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, από τις οποίες προέρχομαι και εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογο για τα ζητήματα αυτά και δυστυχώ διάλογο δεν υπάρχει, τουλάχιστον στο δικό μου τον κλάδο, στη δική μου τη χώρα. Επομένω, κάνω μία έκκληση προ εργοδότε. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε μαζί του, θέλουμε να έχουμε μαζί του τον ανοιχτό διάλογο. Δεν θέλουμε απλώ να διαδηλώνουμε στο δρόμο και αυτό είναι ο μόνο διάβλο επαφή που έχουμε. Ο διάλογος όμως θα πρέπει να λάβει χώρα και σε επίπεδο εταιρεία. Και αυτό Συνήθω δεν συμβαίνει και όταν συμβαίνει είναι ανηλικρινή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνθήκε εργασία στι δικέ μου τι χώρε, στη δική μου τη χώρα, είναι σαφώ κατώτερες από τι συνθήκε εργασία στη Δυτική Ευρώπη και ζητώ την δική σα βοήθεια, τη βοήθεια των Ευρωβουλευτών από τη δική Ευρώπη. Ο κύριο Βάμπ νομίζω ότι θέλει να πάρει το λόγο και νομίζω ότι είναι ο τελευταίος ομιλητή. Είχαμε και ένα νέο αίτημα Μπορείτε όμως να πάρετε παρακαλώ πολύ το λόγο στο επόμενο τμήμα της συζήτησης. Ο κύριε Ρόι θα μιλήσετε στην επόμενη συνεδρίαση. Ο κύριο Φαβ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βρίσκω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το πλαίσιο σήμερα, διότι ε, και οι stakeholders, οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δυνατότητα να συμβάλλουν στη συζήτηση. Ε, όσον αφορά τη συζήτηση στο δεύτερο και στο τρίτο τμήμα τη Στρογγυλής τράπεζα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Όσον αφορά τις τιμές, ε, ε, η κυρία Στάιλερ αναφέρθηκε σε αυτό. Στην περιοχή μου, στο ΚΕΛ, κοντά στο Στρασβούργο, υπάρχει τυπογραφείο που ε, ε, ε, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη διότι πολλοί από τη Γαλλία έρχονται να τυπώσουν τα πράγματα τους εκεί. Νομίζω ότι αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στα διάφορα εμπόδια που δημιουργούνται για το εμπόριο. Νομίζω ότι έχουν να κάνουν και με κάποιες τοπικές παραδόσεις. Επίσης, όσον για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο ε, οι τιμές είναι ψηλότερες από ό,τι σε όλες τις γειτονικές χώρες ε, και ε, κάποιος μου εξήγησε ότι η Auchan έχει το πρόβλημα ότι όλες οι μάρκες, όλα τα προϊόντα μάρκας πρέπει να περάσουν από το Βέλγιο. Εδώ μιλάμε για συμφωνία μεταξύ των λιανοπολιτών. Ε, νομίζω όμως ε, ότι και οι προμηθευτές ε, ευθύνονται για τις διαφορές στις τιμές και πιστεύω ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στο να πει υπάρχουν τεχνητά εμπόδια για τους ε, καταναλωτές ε, στα διάφορα Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες από πού προέρχονται τα διάφορα αυτά εμπόδια. Νομίζω ότι μερικά από αυτά όπως ε, είπατε, μερικά από τα θέματα αυτά αφορούν και το επόμενο τμήμα της συζήτησης, το είπατε και εσείς ο ίδιος. θα ήθελα να καλέσω τώρα τους ομιλητές του πάνελ ε, για δύο λεπτά το πολύ να απαντήσουν ε, στις παρατηρήσεις αυτές, ε, να μοιραστούν μαζί μας τους συλλογισμούς τους. Μήπως κινηθούμε με ανάποδη σειρά, να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Σκίαν και κατόπιν να κλείσουμε με τον καθηγητή κύριο Στυκ. Πολ, έχεις δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, για τα εμπορικά σήματα, το All Brand, καταρχήν μέσω της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου είχαμε τις ίδιες συζητήσεις και τελικά η Γάμα Delta Enterprise ζήτησε μια έκθεση που έχει τώρα 188 σελίδες. Δεν θα σας διαβάσω αλλά η σύνοψη είναι η εξή. Και ακριβώ αυτό το ζήτημα διερευνήθηκε. Την ανάπτυξη τη ίδια ε, του ίδιου εμπορικού σήματο στην Ευρώπη. Ε, το, η σύνοψη είναι ότι η καινοτομία δεν είναι υποπίεση. Ο ρυθμό τη εισαγωγή προϊόντων αυξάνεται. Αυτό ισχύει και για τι βιομηχανικέ μάρκε και για τι ιδιωτικέ ετικέτε. Όμω ε, παραμένει συνεχή η παραγωγή τη βιομηχανική βιομηχανίας ε, τροφίμων. Η μελέτη δεν ε, παρατηρεί πρόβλημα σε σχέση με τις σχέσεις ε, προμηθευτών και λιανεμπόνων στι ιδιωτικέ ετικέτες και μάλλον δεν θα υπάρχει επίπτωση στην καινοτομία σε βιομηχανικό επίπεδο. Ελπίζω να το εγκαταλείψει η ΓΔΕ αυτό το θέμα γιατί είναι πλήρως ό,τι αφορά το πώς ε, βλέπουν οι λιανέμποροι το θέμα αυτό να λαμβάνουν ευθύνη. Αν πιστεύουν ότι οι λιανέμποροι ε, βάζουν προϊόντα με το δικό τους λογότυπο πάνω και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για να εγγυθούν την ασφάλεια, την ποιότητα του προϊόντος κτλ. Δεν ισχύει φυσικά και το κάνουν γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Όπως είπε η κυρία Στάιλερ, είναι η δική του μάρκα. Δεν ε, θα διακινδυνεύσουν το δικό του εμπορικό σήμα και να τελειώσω με κάτι θετικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι κοινά στον ε, τομέα από τους προμηθευτές μέχρι τους λιανεμπόρους και εγώ θα ευχόμουν στην έκθεση που ε, θα προέρθει από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ αλλά και γενικά πολλά από τα θέματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της ε, εσωτερικής αγοράς για όλη την διατροφική λυσίδα να επιληθούν και εσείς ε, συλλογικά να ασκήσετε πίεση στην Κομισιόν για να ε, προφεύγει σε διαδικασίες επί παραβάση. Πολύ ταχύτερα η απάντηση της Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο για, τα μέσα, για τον νόμο για τα μέσα μαζικής ε, ενημέρωσης στην Ουγγαρία δείχνει πόση πίεση έχετε. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και με τις διαδικασίες επί παραβάσης Σας ευχαριστώ. Κατόπιν, ο κύριος Γκαλάσκι. Ευχαριστώ. Θέλω να υποστηρίξω όσα υπόθηκαν από τον Πολ. Στο τέλο, να απαντήσω στην κυρία Στήλερ σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό από την ίδια ετικέτα. Εμεί δεχόμαστε ε, τον ανταγωνισμό από τι ιδιωτικέ ετικέτε. Υπάρχουν ιδιωτικέ ετικέτε που είναι μάλιστα πιο ακριβέ από τα εμπορικά σήματα. Δεν είναι ε, μια κατάσταση άσπρη-μαύρη. Σωσέ πολύ για αυτή την μελέτη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να το διαβάσει κανεί όλη τη μελέτη. Αναφέρθηκε ότι στην ε, Ισπανία η έκθεση αναφέρεται σε σημαντική μείωση αγωγέ νέων προϊόντων, όταν είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι αφορά το μερίδιο στι ετικέτε προϊόντων. σω είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλε θετικέ πτυχέ. Τώρα για την αντιγραφή, το copycat, την αντιγραφή γίνεται και από του λιανεμπόρου, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχουν ε, δύο διαφορέ. Ε, ε, δεν ακούγεται πάρα πολύ ε, για, δεν ακούγεται πάρα πολύ παράπονα κατασκευαστών εμπορικών σημάτων είναι γιατί δεν θέλουν να το δημοσιεύουν πάρα πολύ το ζήτημα. δεν θέλουν να δημοσιεύουν ότι έχουμε αντιγραφή από ένα πελάτη. Επίσης, ε, μια αντιγραφή, ένα copycat ε, μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα στη διαδικασία επειδή ο Λιανέμπορος μπορεί να έχει νωρίτερα πληροφορίες ως πελάτης. Και κάτι ακόμη για τη διαφορά στις τιμές ε, στην ενιαία αγορά. Πράγματι, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς, γιατί εμείς εκπονήσαμε ένα έγγραφο για όσου ενδιαφέρεστε για τους λόγους της διαφορετικότητας των τιμών στην αγορά. Ευχαριστώ να σας το μοιράσουμε. Και όσο είπε και ο Πολ, ε, προηγουμένω. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ε, στη μελέτη τη Κομισιόν ε, τη γάμα δέλτα competition που ξέρουμε πόσο σκληρή στάση κρατεί και η γάμα δέλτα για τα οικονομικά έχουν ζητήσει μια μελέτη για τα θέματα αυτά και τώρα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται υπάρχουν γεγονότα. Η ερώτηση είναι αν έχουμε την ίδια ερμηνεία των γεγονότων. Τώρα, η κυρία Φρούεν. Ευχαριστώ. Όντω είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλες τις παρατηρήσεις που γίνανε. Θα αναφερθώ σε ορισμένες. Ακούστηκε μια παρατήρηση για την αυτορύθμιση. Σίγουρα η προσέγγιση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά την νομοθεσία ή την μη νομοθεσία θα έλεγα, γιατί η αυτορύθμιση έχει λειτουργήσει και λειτουργεί καλά σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ορισμένε περιπτώσει πάλι απαιτείται όμω η νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ακούσαμε, δηλαδή εθνική νομοθεσία σε ορισμένε περιπτώσει, άλλε φορέ ακούμε εκκλήσει για κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις συμβατικές και εμπορικές πρακτικές, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω καθόλου την ε, συζήτηση, η τα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι θέλουμε μία νομοθεσία η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Μία νομοθεσία η οποία θα δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα, γιατί αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ε, τότε δεν έχει και ιδιαίτερη αξία. Να επανέλθω επίσης ε, σε ένα άλλο σημείο. Σήμερα το πρωί είδα στην εργασία μου, στη δουλειά μου, έναν κύριο που εκπροσωπεί μία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ευρώπη και του ζήτησαν να έρθει μαζί μου σήμερα το απόγευμα και μου είπε ότι αφήστε καλύτερα, δεν θα έρθω, θα έρθω όταν συνταξιδοτηθώ. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά καταδεικνύει το πρόβλημα αυτό το οποίο υπάρχει. Ότι οι κατασκευαστές από φόβο δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους υπάρχει ένας φόβος και ο φόβος αυτός υπάρχει ακόμα και για τους μεγάλους κατασκευαστές. Εμείς εκπροσωπούμε και μικρούς και μεγάλους όπως ξέρετε. Υπάρχει λοιπόν ένας διάχυτος φόβος και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε και με τους εκπροσώπους των άλλων ενός που ακούσαμε σήμερα και από κοινού να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ψάχνουμε όλοι κάποια δεδομένα, θέλουμε τα απαραίτητα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια λύση. Όλοι όμως όσοι συμμετέχουμε στην αλυσίδα αυτή του εφοδιασμού θέλουμε να βρεθούν λύσεις και θέλουμε στο τέλος να βοηθήσουμε και τον ίδιο τον καταναλωτή. Κύριε Ντέιβις, σας ευχαριστώ. Πολλά πράγματα ακούστηκαν, καλύφθηκε μεγάλο έδαφος. Όσον αφορά το ζήτημα της συσκευασία, της αντιγραφής, copycat, της ε, ιδιωτικής, ε, του ιδιωτικού εμπορικού σήματος, θα ήθελα να σας παραπέμψω στην έκθεση ΣΥΣΥ για τα παντοπολία, στο παράρτημα 9-10, όπου γίνεται μία αναφορά στο ότι πραγματικά από τη δεκαετία του 1960 και μετά έχουν αυξηθεί τα εμπορικά σήματα, οι ιδιωτικές, τα ιδιωτικά σήματα, σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες των προϊόντων. Και επίσης λέγεται εκεί ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση με την πάρδο του χρόνου μέσα στα πλαίσια της ίδιας κατηγορίας και δίνονται και κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, δίνονται κάποια παραδείγματα για το τυρί τσένταρ ή για κάποιες ε, σημαντικές αλλαγές που γίνανε και οι οποίες οδήγησαν σε πολύ σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το, τα ιδιωτικά σήματα σε άλλα προϊόντα επίσης όπως το γιαούρτι. Και βλέπουμε τελικά ότι υπάρχει μια αρκετά πλούσια και διαφοροποιημένη εικόνα. Και καταλήγουμε τελικά σε έναν κόσμο που υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο που πολλές φορές προκύπτει από το θετικό ουσιαστικά γεγονός ότι έχουμε πολλά προϊόντα ιδιωτικής ε, ετικέτας. Και πολύ συχνά βλέπουμε, αυτό άλλωστε λέει και έρευνα, ότι είναι προϊόντα τα οποία χαίρουν υψηλή εκτίμηση και διατίθενται σε κάποιε χαμηλέ τιμέ. Όσον αφορά το ερώτημα το οποίο ακούστηκε για, την, για το στονισμό CC και FT, καθώ επίση και άλλων οργανισμών που ασχολούνται με τον ανταγωνισμό, υπάρχει συντονισμό κυρίως με άτυπη μορφή, μέσω των Ευρωπαϊκών Δικτύων Ανταγωνισμού και μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΣΑ και μέσω και διμερών επαφών και συνεδριάσεων τόσο των Βρετανικών αρχών στην συγκεκριμένη περίπτωση όσο και άλλων εθνικών αρχών από άλλα κράτη-μέλη όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια βούληση για ανταλλαγή πόρων και ιδεών. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ο, προ... ο καθηγητής Στούκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα με το οποίο ασχολούμαι δεν σχολιάστηκε, ωστόσο θα πω λίγα λόγια, διότι τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δείχνουν ακριβώς τη θέση μου. Πολλά από τα όσα υπόθηκαν, η επιλεκτική διανομή, οι διαφορές στις τιμές, η αγοραστική δύναμη, ε, πολλά από αυτά είναι θέματα ανταγωνισμού και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια του, ε, της νομοθεσίας αντιτράστη. Ε, θα χαρώ πολύ να δω την μελέτη IAA, διότι ε, ε, φαίνεται να υπάρχει, να ετοιμάζεται μια μελέτη που να δείχνει ότι κάνω λάθο. Αν συμβεί αυτό, το θα παραδεχτώ ότι όντω κάνω λάθος, ε, αλλά α περιμένουμε τη μελέτη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή ποικιλία παρεμβάσεων και νομίζω ότι ήταν χρήσιμο που ακούσαμε και από τους ε, λιανοπολιτές αυτοκινήτων, ε, διότι ε, έτσι μας θύμισαν ότι υπάρχουν το μίσο που υπάρχει, υπάρχουν ρυθμίσεις franchising που καλύπτονται από τις γενικές παρεκκλήσεις και ξέρω ότι αρκετοί από τους λιανοπολιτές αυτοκινήτων ανησυχούν που δεν υπάρχει τομεακή ρύθμιση. Ακούσαμε και ε, κάποια πράγματα για εμπορικές πρακτικές που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με τις ε, τιμές. Ακούσαμε θέματα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την καλή λειτουργία της αγοράς. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα τα θέματα αυτά και να ελέγχουμε αν είναι αντίθετα στον ανταγωνισμό. Και αυτό μας θυμίζει τη θέση του κυρίου Στίκ ότι έχουμε το δίκαιο περί ανταγωνισμού. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο ε, τμήμα της συζήτησης όπου θα μιλήσουμε για θέματα προσβασιμότητας στην αγορά. Θα ε, επανέλθουμε σε κάποια από τα εμπόδια που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην αγορά. Και πάλι έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ εμπειρογνωμόνων. Έχουμε την κυρία Πατρίσια Χόκστρατεν που είναι διευθύντρια του FAC Centrum, που είναι ε, μια ένωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της διανομής τροφίμων. Έχουμε τον ε, δόκτορα Reinhard Freicher von ε, Leoprechting. Ζητώ συγγνώμη, ελπίζω να μην κατέστρεψα τελείω το όνομά σας, που είναι μέλος του Συμβουλίου του, της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Ιλιανικής Έχουμε τον Πίτερ Βίλχελμ που είναι γενικός διευθυντής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής ε, ε, Βελγικού Λιανοπολιτή ε, είναι όμως και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Δημόσιες Υποθέσεις. Και τέλος, ε, κάποια που δεν είναι ε, καθόλου ξένη προς την Επιτροπή μας, είναι η πρώτη της εμφάνιση το 2011. Μιλώ για την ε, Μονίκ Γογιένς που είναι Γενική Διευθύντρια της ΜΠΕΟΚ. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χοκ Στράτεν. Πέντε λεπτά. Thank you, Mr. President. Next ναι, ευχαριστώ οι ανεξάρτητοι λιανέμποροι να δέμα τροφίμων δρούν με δικό του κίνδυνο και στις ε, κατοφόρε χρησιμοποιούν ένα είδος μεθόδου έτσι έχετε κατά νου ότι πίσω από τη μεθόδου τη φόρμουλα μπορείτε να βρείτε έναν λιανέμπορο ε, μια μικρή μικρομεσαία επιχείρηση ε, Παραδείγματο χάρη, ε, ε, ε, μπορεί η επιχείρηση αυτή να δραστηριοποιείται στη γειτονιά, να απασχολείται με ειδικέ ανάγκε κτλ. Έτσι φτάνω στο πρώτο συμπέρασμα. Ε, τη στιγμή που οι αρχέ θέλουν να ανοίξουν την προσβασιμότητα στην αγορά, στην πόλη του θα πρέπει να εμπλέξουν και του τοπικού επιχειρηματίε στα σχέδιά του, καθώ υπάρχει προστιθέμενη κοινωνική αξία. Είναι πολύ σημαντικό Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες διέξοδοι. Οι δικτές και ε, όσοι αναπτύσσουν τις, την ιδιοκτησία δεν ε, λαμβάνουν υπόψη τους ανεξάρτητους επιχειρηματίες και έρχομαι τώρα στο δεύτερο συμπέρασμα ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στις νέες αγορές και να αποκτούν διεξόδους για τα αγαθά δικές τους ε, ε, και θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις αρχές. Ε, είναι ε, πάρα πολύ σημαντική και είναι εξάρτητη η χρηματοδότηση ως εργαλείο για την ε, προσβασιμότητα στην αγορά. Λόγω της ε, κρίσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, έχουν περιέλθει σε δύσκολη θέση. Πρέπει όμως να σταματήσουν να ζητούν οι τράπεζες τις εγγύσεις, γιατί οι εγγύησεις ε, που υπό τον κανονισμό 330 του 2010 μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αυστηρές υποχρεώσεις στον ανεξάρτητο λιανέμπορο και σε όλους τους ανεξάρτητους λιανέμπορους. Ε, χρειάζεται καλές συμβάσεις που πρέπει να ξεκινάνε από ένα προσυμβασιακό στάδιο. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να λαμβάνει ορθές πληροφορίες. Αυτή η προσυμβατική φάση δεν ρυθμίζεται στις κατοχώρες ε, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα στην Γαλλία και στο Βέλγιο που θα ήταν καλό να τα ακολουθήσουμε. Κατόπιν έχουμε συμβάσει δικαιοκρισία με υποχρέωση ε, αυτός που αναλαμβάνει δικαιοκρισία να ε, προσφέρει στον εταίρο του το, το κατάστημά του σε μια ανταγωνιστική τιμή στο τέλος. Αυτό θεωρείται από τις αρχές ότι παρεμποδίζει τον ελευθερό ανταγωνισμό. Το συμπέρασμά μου είναι ότι θα έπρεπε να άρουμε τις ρήτρε του μη ανταγωνισμού στο τέλος των όρων. Θα πρέπει να καταργήσουμε την υποχρέωση της πώληση του καταστήματος σε μη ανταγωνιστική τιμή και θα πρέπει να ρυθμίσουμε το προσυμβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και εδώ η Κομισιόν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρόσθετοι όροι πρέπει να καθορίζονται προκειμένου να διασφαλίσουμε το θεμητό ανταγωνισμό, ιδίω ε, αν ε, ο προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα καταναλωτών. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να αποφύγουμε τον κανιβαλισμό της επικράτειας του ανεξάρτητου λιανεμπόρου από τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου ε, του franchiser σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στην αγορά και την απορρίθμιση, πρέπει να πω ότι θα πρέπει να θέσουμε σε μια σειρά τους κανόνες. Ε, όμως πρέπει ε, να γνωρίζει η αγορά τι θα ωφελήσει και τι θα ωφελήσει τους ανεξάρτητους λιονεμπόρους. Δηλαδή, ε, το να απορριθμίζουμε... Ε, τους κανόνες θα μπορούσε να ωφελήσει πολλούς καταναλωτές αλλά και λιανεμπόρους. Και ας έρθω στο τελικό συμπέρασμα ε, που είναι ε, το εξής, ότι αν υπάρχει μια ελεύθερη αγορά για ανεμπόρων, τότε ο καταναλωτής θα μπορούσε ε, να επιλέξει μεταξύ των ε, πολυκαταστημάτων, των πολυεθνικών έτσι λοιπόν θα πρέπει ε, τα ευρωπαϊκά όργανα να δημιουργήσουν ίσους κανόνες προκειμένου να δώσουν σε όλες τις μορφές λιανικής τις αναγκαίες ανταγωνιστικές ευκαιρίες και χρειαζόμαστε γι' αυτό κάποια υποστήριξη ε, για τους ε, λιανεμπόρους ε, όταν μιλάμε για μικρές και μισές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, σας ευχαριστούμε για τη παρουσίασή σας και σας ευχαριστούμε και που σεβαστήκατε το χρόνο. Κατόπιν έχουμε τον κύριο Ράιντχαρτ. Ναι, περιμένω τις διαφάνειες μου καταρχήν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο τίτλος ε, της ε, συζήτησης, το άνοιγμα της αγοράς δηλαδή για επιχειρήσεις και καταναλωτές, είναι πολύ καλός τίτλος διότι αυτό είναι ε, το θέμα που αφορά το μισό δισεκατομμύριο καταναλωτών και τα 6 εκατομμύρια επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική έκθεση εξετάζει τον ε, τομέα της λιανικής στην Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά ε, και Επίσης ε, περιμένουμε και την ε, έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας εξετάσουμε λοιπόν ε, τον ρόλο κλειδί του εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία. Καταρχήν να εξετάσουμε τη σχέση εμπόριο-καταναλωτής. Ο ρόλος αυτός αφενός επηρεάζεται από την σχέση με τον παραγωγό ε, από την άλλη ε, έχουμε τους όρους των συμβάσεων και τη διαμόρφωση των τιμών και οι δύο πλευρές εξαρτώνται η μία από την άλλη και έτσι υπάρχει ισορροπία. Γι' αυτό απορρίπτουμε προσπάθειες ε, με νόμους ή με κώδικες δεοντολογίας να επηρεαστεί η σχέση αυτή τέτοιοι κανόνες οδηγούν σε στρέβλωση της, ε, του ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ε, συμφωνήσω με την έκκληση της κυρίας Μπίλτ και του κυρίου Σβάπ. Θα εξετάσουμε λοιπόν ποιες ε, συμπεριφορές θεωρούμε προβληματικές. Ας εξετάσουμε την άλλη άκρη της αλυσίδας, τους καταναλωτές δηλαδή. Και θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στην ίδια μελέτη το παρακολούθηση αγοράς. Ε, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε προϊόντα από άλλα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες και έτσι υποφελούνται από την ε, ενιαία αγορά. Ε, Ε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, 30.000 ε, εργαζόμενοι στο ευρωπαϊκό λιανικό εμπόριο, το οποίο σημαίνει ότι μία σε επτά θέσεις εργασίας της Ευρώπης ε, βρίσκεται στον τομέα του εμπορίου. στην ε, προσπάθεια δημιουργίας ε, μιας ε, βιώσιμης οικονομίας η αλυσίδα προμήθειας παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης το εμπόριο έχει το ρόλο διασφάλισης ε, της πρόσβασης σε προϊόντα καλή τιμής ε, για τους καταναλωτές. Ε, περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το εμπόριο είναι το κλειδί της ενιαίας αγοράς και αποτελεί την πύλη του καταναλωτή στον κόσμο των προϊόντων. Αυτή η απλή σχέση όμως μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η εσωτερική αγορά της Ευρώπης εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει σαφή υποχρέωση να εξαλείψει τα εμπόδια ε, που εμποδίζουν την ε, πρόσβαση στην ενιαία αγορά στις ε, επιχειρήσεις. Βασικός τομέας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η εσωτερική αγορά. Πολλοί άνθρωποι ξεχνάνε ότι οι συνέπειες αυτές είναι ε, ε, οι θετικές συνέπειες είναι μετρήσιμες και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 2,5 ε, εκατομμύρια επιπλέον θέσεων απασχόλησης δημιουργήθηκαν με την εξάλληψη των εμποδίων στο εμπόριο, αλλά μας απειλεί ένας κίνδυνος ε, σε κάποια ανατολικά κράτη-μέλη υπάρχουν κάποιοι προβληματικοί κανόνες ε, που ισχύουν και σε άλλες ε, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις από άλλα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν κάποιες προβληματικές ε, συμφωνίες, ε, υπάρχουν κάποιες, κάποιοι κανόνες που δημιουργούν διακρίσεις και που παραβιάζουν τις βασικές ελευθερίες που εγγυάται η συνθήκη. Και περνάμε στην τελευταία διαφάνεια, πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε ένα παράδειγμα από την Ουγγαρία. Με την δημιουργία ενός αναδρομικού φόρου, οι εσωτερικές επιχειρήσεις εξαιρέθηκαν από την ε, υποχρέωση υποβολής του φόρου αυτού. Αυτό ή αποτελεί ε, κατάφορη διάκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βίλχελμ. Um, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν με παρουσιάσατε, είπατε βέβαια ποιος είμαι. Είμαι πρόεδρος μιας εταιρείας η οποία εκπροσωπεί εμπορικά κέντρα τόσο στο Βέλγιο όσο και σε άλλες χώρες και μιλώ βέβαια εδώ πέρα ως εκπρόσωπος κυρίως του ICSC, του Διεθνού Συμβουλίου Εμπορικών Κέντρων. Μου ζητήσετε να απαντήσω στο εξή ερώτημα. Υπάρχουν κάποιε προτάσει ή λύσει προκειμένου να αυξηθεί η ελεύθερη πρόσβαση των λιανοπολιτών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οποιοδήποτε έχει πάει σε εμπορικό κέντρο θα έχει συνειδητοποιήσει ότι εμπορικά κέντρα συνήθω απαρτίζονται από πολλού διεθνεί λιανοπολιτέ. Τα εμπορικά κέντρα λοιπόν εξορισμού απαντούν, αν θέλετε, στο ερώτημα αυτό. Βέβαια, ξέρετε ότι συχνά επικρίνονται τα εμπορικά κέντρα γιατί ε, υποτίθεται ότι σκοτώνουν τον τοπικό μικρό πολιτή και γι' αυτό το λόγο απαγορεύονται σε ορισμένες πόλεις, τουλάχιστον από το κέντρο των πόλεων. Επομένως το ερώτημα είναι το ακόλουθο. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα εμπορικά κέντρα ή όχι. Εγώ θα προ... απαντώντας στο ερώτημα αυτό θα απαντήσω και στη δική σα την ερώτηση για την προσβασιμότητα στην αγορά λιανικής πώληση. Το πιο σημαντικό για να λέμε πολιτή είναι η τοποθεσία. Και όταν λέω τοποθεσία αναφέρομαι σε ένα μέρος όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περνάνε, όπου μπορούν πάρα πολλοί να δουν τη βιτρίνα του καταστηματάρχη κτλ. Τι είναι ένα εμπορικό κέντρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πούνε ότι είναι ένας χώρος φτιαγμένος από γελί με πάρα πολλά καταστήματα που έχει και πάρκινγκ. Βέβαια για μας αυτό δεν αποτελεί ορισμό. Ένα εμπορικό κέντρο για μας είναι ε, ο συνδυασμός ε, ορισμένων ε, καταστηματαρχών που έχουν αγοράσει ή έχουν νοικιάσει συγκεκριμένον χώρο και συνδυάζεται αυτό με μια σημαντική μάζα πελατών. Επίση, πρέπει να σα πω ότι όταν λέμε σημαντική μάζα, κριτική μάζα, εννοούμε ότι υπάρχει ο απαραίτητο αυτό όγκο, η απαραίτητη επιφάνεια που επιτρέπει την παρουσία πολλών διαφορετικών μαρκών. Ποια υπάρχουν κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά όσον αφορά το εμπορικό κέντρο, τα εμπορικά κέντρα. Τα εμπορικά κέντρα σκοτώνουν ουσιαστικά τον μικρό πολιτή. Στο, στο Βέλγιο θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έχουμε ένα νέο εμπορικό κέντρο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε μια νέα πόλη που λέγεται Λουβέο Λανέβ η πόλη αυτή δεν παρουσίαζε κάποια σημαντική ανάπτυξη και είπαμε στις τοπικές εθνικές αρχές ότι αν δημιουργεί το ένα εμπορικό κέντρο θα αυξανόταν πολύ περισσότερο η πόλη και θα υπήρχε και μια πιο έντονη τόνωση αν θέλετε του κοινωνικού ιστού και οικονομικού ιστού στις, στην πόλη αυτή. Και αυτό ακριβώ συνέβη. Κατασκευάστηκε το εμπορικό κέντρο και η Λουβένα Λανέβ έπαψε να είναι απλώ μια πόλη κοντά στο πανεπιστήμιο και έγινε μια πραγματική πόλη. Τώρα, ε, επανερχόμενο πάλι στο ερώτημα αυτόν, τα εμπορικά κέντρα καταστρέφουν τον ε, μικρό Ελληνοπολιτή. Δεν θα ήθελα να επισέλθω πάλι σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείτε να αποφύγετε την παρουσία των εμπορικών κέντρων, καθώ επίσης και τον ενδιαφέρον που δείχνουν οι πελάτες. Στο κέντρο τη Διαγής δημιουργήθηκε ένα εμπορικό κέντρο, όπου ε, Είχαμε το πρώτο Prime Mart, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Βρετανοί κάτοικοι του Βελγίου. Είχαμε επομένω πάρα πολλού πελάτε οι οποίοι ερχόντουσαν ακριβώ στο κέντρο τη Λιέγη, ακριβώ για να πάνε στο κατάστημα αυτό που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πολύ συχνά οι μεγάλες εμπορικές μάρκε λειτουργούν μέσω ενό συστήματο franchising, δικαιοχρησίας. Κατά αυτόν τον τρόπο ο πελάτης καταφέρνει να έχει πρόσβαση στα προϊόντα αυτά. Στα δύο αυτά μεγάλα εμπορικά κέντρα στα οποία αναφέρθηκα με διασύτε υπάρχουν πάρα πολλοί επιμέρους λιανοπολιτές οι οποίοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εμπορικά κέντρα. Ουσιαστικά όμω αυτοί που κινούν την αγορά είναι οι μικροί λιανοπολιτέ. Μπορεί να εκπροσωπούν μια μεγάλη εταιρεία, αλλά ουσιαστικά αυτοί στο δικό του επίπεδο καταφέρουν να κινήσουν περισσότερο την αγορά. Θα μπορούσα να σας δώσω και παραδείγματα άλλων πολιτών όπου μπορούν να κατέχουν μια μικρή επιφάνεια στο εμπορικό κέντρο. παρόλα αυτά ο κύκλος εργασιών τους είναι διπλάσιος ή πολύ μεγαλύτερος από άλλα μεγαλύτερα καταστήματα. Επίσης τους κεντρικούς ε, εμπορικούς ε, δρόμους βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τα νίκια τα οποία πολύ συχνά μπορεί να είναι ακριβά. Το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίζεται στα εμπορικά κέντρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο κύκλος εργασιών. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι ε, υπάρχουν κάποιες μεγάλες εταιρείες οι οποίες εκειώνται χαμηλά ενίκια για την παρουσία τους στα εμπορικά κέντρα και αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους μικρούς λιανοπολίτες. Ένα ακόμα ερώτημα. Αληθεύει ότι τα εμπορικά κέντρα επιβάλλουν πολύ μεγαλύτερους φόρους εξυπηρέτησης από ό,τι τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν κερδοφορούμε, δεν δημιουργούμε κέρδη μέσω των τελών, αν θέλετε, εξυπηρέτησης. Θα μπορούσατε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας τα όσα σας είπα και θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε και στην εφαρμογή την μεγαλύτερη υλοποίηση εμπορικών κέντρων και θα μπορούσατε να το κάνατε αυτό υποχρεώντας τα κράτη-μέλη εκείνα τα, να, τα οποία δεν εφαρμόζουν την ε, την οδηγία για τις υπηρεσίες να αρχίσουν να την εφαρμόζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη όπως στη Γαλλία όπου γίνονται κάποιες προσπάθειες παράκαμψης της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πολλές φορές κάποιοι οργανισμοί αλλάζουν το όνομά τους, αλλά τελικό του στόχος τελικά είναι να παρακάμψουν την οδηγία για τις υπηρεσίες και κατά αυτόν τον τρόπο στρεβλώνουν τον αγωνισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα όσα είπατε είναι πολύ σημαντικά για το ζήτημα της ανεξαρτησίας Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Μονίκ Γκογιένς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κορατσαβίλτ. Εγώ θα σας ε, παρουσιάσω τη σκοπιά των ε, καταναλωτών, ε, αλλά δεν θα το κάνω από την τοπική αστική σκοπιά. Μέσα σε πέντε λεπτά θέλω να σας αναφέρω πάρα πολλές προκλήσεις, αλλά θέλω να προσπαθήσω να αυτορυθμιστώ προς το χρόνο μου Πρόεδρε, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε κάπως διστακτικοί ε, για το θέμα της αυτορύθμισης, έτσι παρακολουθήστε με παρακαλώ και ε, φροντίστε να μην ξεπεράσετε το χρόνο που έχουμε συμφωνήσει. Θέλω να αφαιρθώ στην πληροφορία στους καταναλωτές, στην ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στην πρόσβαση των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, λειτουργία, αγορά πνευματικά, αν ε, είναι ενημερωμένο σωστά ο καταναλωτή και μπορεί να επιλέξει στο πλαίσιο αυτό θέλω να θέσω τρία ζητήματα. Καταρχήν, υπάρχει προ στιγμή μία τάση να, μπαίνουν, να ε, χρησιμοποιούμε εργαλεία συγκρίση των τιμών και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η επιλογή των καταναλωτών δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή. Δηλαδή, ε, ε, δίνεται μία σημασία στην τιμή αλλά πρέπει να την εντάξετε σε αυτή την προοπτική και επίσης οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εξαντλητικές δηλαδή να καλύπτουν όλη την αγορά θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένε, ε, δηλαδή να επικαιροποιούνται συχνά για τις τιμές που προτείνονται από τους διάφορους προμηθευτές και θα πρέπει να είναι και ακριβείς. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πλήρες, να μην ξεχνάμε τους φόρους ε, ή οτιδήποτε άλλο προστίθεται στην αρχική τιμή και θα πρέπει να έχουμε και ανεξάρτητες πληροφορίες, δηλαδή ε, ε, κάτι ακόμη που θέλω να πω έχει να κάνει με τις ιδιωτικέ ετικέτες. Πρέπει να αντιδράσω στην παρέμβαση του Ιταλού συναδέλφου. Θέλω κάποιος να το πει γιατί δεν είναι εδώ. Εμείς ως καταναλωτές πιστεύουμε ότι οι ιδιωτικέ ετικέτες, για τις ιδιωτικέ ετικέτες οι ναι, μπορεί παίρνουν την ευθύνη έναντι των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό για τον καταναλωτή να το ξέρει αυτό. Και θέλω να είμαι κάπως προκλητική αν μου επιτρέπετε γιατί για τα προϊόντα ο καταναλωτή ε, δεν έχει απαραίτητε πληροφορίε για το ποιο το παράγει. Αν έχουμε παραδείγματο χάρη μία μάρκα από γιαούρτι, ξέρουμε ποιο επεξεργάζεται το γιαούρτι, αλλά δεν ξέρουμε πού προέρχεται το γάλα, ούτε ξέρουμε ποιο ε, ταίζει την Αγελάδα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι ο βασικό παραγωγό, αν θέλετε να αναφερθούμε στην ποιότητα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να μην κάνουμε τεχνητέ ε, Διακρίσει μεταξύ των, ιδιωτικών ετικετών και των ε, ε, προϊόντων με εμπορικό σήμα. Δεύτερον, πρόσβαση των καταναλωτών στην αγορά και στα αγαθά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέλουμε να έχουμε μια θεμητή αγορά, να μην υπόκεινται σε εισαγωγή διακρίσεων καταναλωτέ. καταναλωτές ε, βάσει της επικράτεια. Και αυτό συμβαίνει ακόμη στην Ευρώπη. Αν προσπαθεί να αγοράσει στην Μαδρίτη με την πιστοτική του κάρτα ειστήρια για το μετρό, δεν μπορεί να τα πάρει αυτά στο αεροδρόμιο ε, με την πιστοτική του κάρτα και μπορείτε να δείτε ότι οι ξένες πιστοτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές από αυτά τα μηχανήματα. Ενώ ε, εκεί πρέπει να εξυπηρετούνται οι ξένοι ταξιδιώτε. Όμω τελικά οι κάρτε του δεν ε, γίνονται αποδεκτέ. Ε, οι καταναλωτέ βλέπουν πολύ μεγάλη άρνηση παράδοση, παραδείγματο χάρη όταν ψωνίζουν από ιστοσελίδε. Και πολλέ φορέ δεν μπορούν να μπουν σε μια ξένη ιστοσελίδα γιατί συστηματικά και αυτόματα ξανά οδηγούνται στην ιστοσελίδα την εγχώρια τη εταιρεία βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, κάποιοι πρακτικοί περιορισμοί για την ε, επιλεκτική διανομή, όμως ε, δεν ανοίγει επαρκώς η αγορά και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μάλλον αυτή η ρήτρα που επιβάλλεται για το ηλεκτρονικό εμπόριο κλείνει την αγορά αν θέλει να αγορασει καποιο κάποιος ε, ένα MP3 ε, στη Γερμανία ε, πρέπει να πληρώσει 2,56 ευρώ ενώ στην Ευστρία από 13 22 ευρώ ε, Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι φόροι για το copyright διαφέρουν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική τιμελόγηση και επομένω μπορεί να μην έχουν πρόσβαση καταναλωτές στα αγαθά. Κάτι ακόμη, προκειμένου να έχουμε μια θεμητή αγορά, πρέπει να παρέχονται στου καταναλωτέ οι λόγοι για να έχει εμπιστοσύνη. Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Προς στιγμή οι πληρωμέ στο διαδίκτυο επικεντρώνονται πάρα πολύ στι πιστοτικέ κάρτε, ενώ υπάρχουν και άλλα μέσα πληρωμή που θα μπορούσαν να είναι πιο ασφαλείς για του καταναλωτέ, Έχουμε ανησυχίε για την ιδιωτικότητα και καλωσορίζουμε ε, την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο μοντέλο για το σημερινό καταναλωτή και θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή ΙΜΚΟ να μην χάσει την ευκαιρία να παράσχει στους καταναλωτές μια θεμητή προστασία όταν μιλάμε για τα ψηφιακά προϊόντα. Γιατί ξέρουμε ότι θα ψηφιστεί σε λίγες ημέρες ε, ε, το σχετικό νομοθέτημα και έτσι λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και Επίσης ε, χρειαζόμαστε δικαιώματα ε, για τους καταναλωτές που να ισχύουν σε όλη την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ισχύουν και στην πραγματική ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, σαφή παρουσίαση και ευχαριστώ που πήρες και την ευκαιρία να καλύψεις και θέματα που αφορούν την αυριανή μας συζήτηση για τα δικαιώματα των θα δώσω τώρα την Προεδρία στην κυρία Κορέτσα Μπίλτ για μισή ώρα, γιατί ε, πρέπει να μεταβώ σε άλλη συνεδρίαση και εκεί θα συμμετέχουν ε, και ψηφοφόροι από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε δεν έχω την πείρα του μάλκον στην Προεδρία. Έχω όμως ένα εξαιρετικό κατάλογο μιλητών και θα ήθελα να ε, ξεκινήσω με τον Γιώσεφ Όργανας Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Από τη Σλοβακία παρακαλώ έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Στείλαμε εγκαίρως στην Επιτροπή τη δήλωσή μας, ε, καθώς και στην κυρία Κορατσαπίλ, ε, γι' αυτό κάποιες παρατηρήσεις. Ε, η Σλοβακική και η Τσεχική Ένωση Εμπόρων επικροτούν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι στιγμής όμως η έκθεση δεν προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις. Καταρχήν ε, θα πρέπει ε, σε όλο το έγγραφο να χρησιμοποιούμε την ε, ίδια οικονομική ορολογία και να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε οικονομικούς όρους. Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να μην υιοθετηθεί νομοθεσία στην Ευρώπη που να προκαλεί διακρίσεις. Για παράδειγμα, ανάμεσα στην Τσεχία και την Σλοβακία και οι δύο χώρες ε, προσέφηγαν στην Κομισιόν χωρίς να έχουν λάβει καμία οριστική θέση μέχρι σήμερα. Όσον αφορά το τμήμα 6, παρατηρούμε ότι η διατύπωση του θέματος αυτού ε, υπερασπίζεται την ε, μεγαλύτερη παραγωγικότητα του τομέα. Στο σημείο 2, 1, 2, 3 εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, κανόνες ε, για την καλύτερη τήρηση των ε, προθεσμιών για την εξόφληση τιμολογίων. Στα συμπεράσματα λέει ότι υπάρχει μια έλλειψη νομοθεσίας, ωστόσο τίθεται το θέμα της επιβολής των σχετικών νόμων και θα παρακαλούσαμε την Κομισιόν να ακολουθήσει τη στάση μας. Ευχαριστώ. Ε, από ό,τι κατάλαβα μιλάτε εκ μέρους ε, και της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Ε, μήπως ο κύριος Τεβέρα θέλει να πάρει το λόγο ή αν καλυφθήκατε. Ε, έπρεπε να αποχωρήσει. Ωραία. Προχωρώ στον επόμενο μιλητή. Μάουριτς Ρούκε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η οργάνωσή μου ε, βλέπει αισιόδοξα την γενική σας προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη πολλούς διάφορους ε, πολιτικούς στόχους. Θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε σε δύο ερωτήσεις. Οι άμεσες πωλήσει ε, αντιπροσωπεύουν 10 εκατομμύρια ανεξάρτητων πολιτών στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι γυναίκες. Δεν Πρόκειται για ε, πλήρη απασχόληση και αυτό καθιστά δύσκολη την ε, ρύθμιση του τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς η Επιτροπή, εσείς η εισηγήτρια, ε, έχετε σκοπό να συμπεριλάβετε το καθεστώς αυτών στην έκθεσή σας και δεύτερον ε, πόσο, ε, πόσα είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε για τις γυναίκες ε, και το επιχειρηματικό πνεύμα. Θα δώσω δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή να απαντήσει μετά. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Χένρικ Φανόστρομ. Ζητώ συγγνώμη αν δεν προφέρω σωστά στα Ολλανδικά το όνομά σας από τον ε, από την Ολλανδική Ένωση Ιλιανικής Πόλησης. Ευχαριστώ πολύ κυρία κορατσαπίλτ, Η κυρία Κόιενς ε, αναφέρθηκε στην, ε, στις εδαφικές διακρίσεις και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τους περιορισμούς στις προμήθειες. Να επανέλθω στο προηγούμενο πάνελ. Ο κύριος Ντέιβις από την Βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού είπε ότι το θέμα δεν είναι βρίσκεται ανάμεσα στους ε, μεγάλους λιανοπολιτές και στις ε, μεγάλες μάρκες. Ε, εγώ διαφωνώ. Η μεγάλες ενώσεις αγοραστών δεν έχουν την δύναμη να ορίσουν τις τιμές. οι κατασκευαστές ε, ε, αναγκάζουν τις ε, αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αγοράσουν τα προϊόντα από τις θηγατρικές τους εταιρείες. Αυτό μπορεί να είναι έξυπνο από πλευράς των μεγάλων επιχειρήσεων αυτών που πουλούν προϊόντα μάρκας, αλλά δεν επιτρέπουν στα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν διασυνοριακά ώστε να πετύχουν τις καλύτερες τιμές. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στα ε, Ολλανδικά σούπερ μάρκετ και στους ε, πελάτες τους. 350 ε, εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να γλιτώσουν τα Ολλανδικά σούπερ μάρκετ, ισχυρίζονται, αν θα μπορούσαν να αγοράσουν τα προϊόντα αυτά από το εξωτερικό. Και θα ήθελα κλείνοντα να πω ότι θα ήταν πολύ καλό και για το σούπερ μάρκετ και για του πελάτε του, εάν εσεί, τα μέλη τη Επιτροπή ΙΜΚΟ, ε, καταφέρουν να είναι ε, ελεύθερη επιλογή από πού θα αγοράσουν τα προϊόντα ε, μάρκα εντό Ευρωπαϊκή Ένωσης σε το σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χοϊσμάν, παρακαλώ. Η κυρία Χοϊσμάν, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε που μα δίνετε τη δυνατότητα μέσω τη επικοδομητική αυτή πλατφόρμα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καταρχά, θα ήθελα να υποστηρίξω τα όσα υπόθηκαν πριν από λίγο για την ε, απουσία εσωτερική αγορά και εμεί ε, ουσιαστικά έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε κάποια εμπόδια τα οποία υπάρχουν στην εσωτερική αγορά και καταλήγουμε κατά αυτόν τον τρόπο και στο θέμα της ε, σημερινής μας συζήτησης, δηλαδή ότι θα πρέπει να δίνουμε στους καταναλωτές πρόσβαση στα προϊόντα. Ένα από τα εμπόδια τα οποία εντοπίσαμε είναι για παράδειγμα η δυνατότητα του καταναλωτή να έχει έγκαιρη και γρήγορη πρόσβαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα. Και αυτό ουσιαστικά προβλέπεται στο νέο κανονισμό για τα καινοτόμα τρόφιμα, το οποίο βρίσκεται σε φάση συνδιαραγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι ε, ένα καινοτόμο προϊόν θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν τα επίπεδα χολυστερίνης. Χρειάστηκε τρία χρόνια να περάσουν προκειμένου το προϊόν αυτό να διατεθεί στην αγορά και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ωφελεί τον καταναλωτή. Όλα λοιπόν αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις Υπάρχει και το ζήτημα αυτό της εξέβρασης των πόρων για τους λιανοπολιτές και εμείς συμφωνούμε μαζί τους ότι θα πρέπει να έχουμε μία καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τους καταναλωτές, το περιβάλλον, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, για να απευθυνθώ και στην Μονίκ, στα όσα είπε δηλαδή για την πληροφόρηση, σαφώς συμφωνούμε με τους ε, στόχους της ΜΠΕΟΚ όσον αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών ε, Για τα προϊόντα εμπορικού σήματος εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο να υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά. Το θέμα όμω είναι πόσες πληροφορίες έχουμε, πού και με ποια μορφή, πώς μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες με ηλεκτρονικό τρόπο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές οι οποίοι θέλουν διαφορετική πληροφόρηση. Άλλοι επιθυμούν να έχουν περιβαλλοντικέ πληροφορίε, άλλοι θέλουν διατροφικέ πληροφορίε, άλλοι θέλουν πληροφορίε όσον αφορά τη σύσταση και την προέλευση του προϊόντο. Χρειάζεται λοιπόν να αποκριθούμε σε όλε αυτέ τι ανάγκε και αυτό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε είναι θένε στην ετικέτα όλε αυτέ τι πληροφορίε. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Σε ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πολύ όλου για τι παρεμβάσει σα. Μπορούμε τώρα να δώσουμε τα... το λόγο στον κύριο Βάιγκα από την Παγκόσμια Οργάνωση Ελληνικής Πώλησης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ περίπου ένα εκατομμύριο μικροεπιχειρήσεις, είναι μικροπολιτές στην Ευρώπη Άκουσα λοιπόν όλες αυτές τις παρατηρήσεις που γίνανε για την ανεξαρτησία, πώς μπορεί κανείς να κινηθεί ως πολιτής ανεξάρτητα τόσο στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους όσο και στα εμπορικά κέντρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν να εξελιχθούν οι μικροπολιτές αυτοί με τρόπο ανεξάρτητο στα πλαίσια της λιανικής αγοράς και πώς θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να αυξήσουν ουσιαστικά το μέγεθός τους και την παρουσία τους και πώς μπορούν να καταλήξουν να γίνουν μεγάλες μάρκες όπως τα σούπερ μάρκετ Tesco και το κατάστημα Marks Spencer. Αναφερθήκατε επίσης στην ασφάλεια των τροφίμων, στην τοπική παραγωγή των τροφίμων και Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η απαραίτητη προσβασιμότητα από τους μικροπολιτές αυτούς οι οποίοι θέλουν να αναπτυχθούν και σε νέες αγορές. Πρέπει ακριβώς να τους δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και σε άλλες χώρες και να φέρουμε σε μια πραγματική ευκαιρία που θα πρέπει να τους δώσουμε όχι μόνο θεωρητικά και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στην πράξη θα πρέπει οι ε, μικρές αυτές επιχειρήσεις, οι μικροπολιτές να μπορούν ε, να αναπτυχθούν επιχειρησιακά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάλι με την ίδια σειρά θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές. Σας ξεκινήσουμε από την Πατρίσια Χόγκστράτεν, από τη Βακ Κέστρομ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε θερμηνία στα Ολλανδικά, επομένως αποφελούμε τις ευκαιρίες να μιλήσω τη γλώσσα μου, λέει ομιλήτρια. Μπορείτε να μιλήσετε Ολλανδικά, λέει η Πρόεδρος. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Βίλχεμ, ο οποίος είπε ότι ε, όσοι ε, δραστηριοποιούνται στα πλαίσια δικαιοχρησίας έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στα πλαίσια εμπορικών κέντρων από ότι αν έχουν ε, δικά τους ανεξάρτητα καταστήματα. Οι άνθρωποι αυτοί μέσω αυτής της αυτορύθμισης έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν οι ίδιοι τη σύμβαση στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιούνται και έχουν επίσης και τη δυνατότητα να μην ανανεώσουν τη σύμβαση αυτή μετά από μερικά χρόνια. Ίσως για αυτό το λόγο ορισμένες μεγάλες εταιρείε, ορισμένοι σημαντικοί παραγωγοί δεν θέλουν να δώσουν συμβάσεις στους ανθρώπους αυτούς. Όσον αφορά τώρα τους ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, ε, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι προβλέπει η νομοθεσία των 27 κρατών μελών για αυτούς. Ιδίως όταν ε, έχουμε να κάνουμε με ε, τα καταστήματα ηλεκτρονικών συσκευών. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε περισσότερο μία ένα καλύτερο σύστημα ηλεκτρονικής πώληση και θα πρέπει ένας καταναλωτής, για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να αγοράσει από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν στην ε, χώρα αυτή. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάμε για 27 κράτη-μέλη. Υπάρχει και το ζήτημα βέβαια της ε, διανομής της προμήθειας. Οι ε, προμηθευτές δεσμεύονται από την ε, εθνική τους νομοθεσία σε κάθε περίπτωση, την τοποθεσία, δηλαδή την νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη και νομίζω θα πρέπει να ληφθεί μια λύση για το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Ράνιχαρτ Φράιερ Βον Λέομπρέχτινγκ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική περιοχή στον κόσμο, τότε χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Ανάπτυξη πετυχαίνουμε με τις επενδύσεις. Επενδύσεις ε, θα πετύχουμε εάν οι επιχειρήσεις έχουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο, το οποίο δημιουργείται με τη σειρά του από την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό οι διάφοροι παράγοντες στην οικονομία θα πρέπει να δημιουργήσουν αυτή την οικονομία, ώστε όπου τελικά η νομοθεσία είναι το έσχατο μέσο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ε, για να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε. Γι' αυτό είμαι ε, υπερασπιστής ε, της πλήρους εναρμόνισης. Η εμπιστοσύνη όμως είναι και η προϋπόθεση για να μπορούμε εμείς ως μεμονωμένοι έμποροι να ε, εργαζόμαστε αποτελεσματικά, διότι όταν επανέλθει ο ίδιο πελάτη, ε, σημαίνει ότι θα έχουμε κάνει καλά την ε, δουλειά μας. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την κυρία Γκογέν. Θα πρέπει να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες ώστε να μπορούν να ε, επωφεληθούν ε, από τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Ε, δεν είμαι βέβαιος αν η συσκευασία είναι ο μόνος τρόπος να παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πιστεύω ότι πάντως θα πρέπει να επιτρέψουμε στον πελάτη να έχει το, τις, τους σωστούς τρόπους πληροφόρηση ώστε να λάβει σωστή και εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με τις αγορές του. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελεσματικό ε, και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Microphone, please. Θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου, αν δεν σας πειράζει. Θα μιλήσω γαλλικά. Θέλω να αντιδράσω στα όσα άκουσα μόλις. Ε, είναι διαφυσβήτητο ότι η κριτική που γίνεται στο εμπορικό κέντρο είναι ότι είναι αντιγραφή το ένα του άλλου και έχουμε παντού το ίδιο μοντέλο και τις ίδιες μάρκες. Ε, όμως ε, για μας ήταν σημαντικό να έχουμε ένα συνδυασμό διεθνών εμπορικών σημάτων αλλά και ανεξάρτητων εμπόρων στα εμπορικά κέντρα είναι πιο εύκολο να ευνοήσουμε την έλευση ε, διεθνών ε, εμπορικών σημάτων ε, από ό,τι στους κυρίους δρόμους, στους κυρίους εμπορικούς δρόμους, γιατί εκεί κάποιος πρέπει να μπορεί να δώσει πολλά χρήματα για να έχει ένα κατάστημα και δεν, το έχουν οι δεν την έχουν οι μικροί αυτή τη δυνατότητα. Έτσι λοιπόν προκειμένου ε, αυτή η μάλλον ε, που εμποδίζουν ε, τους μικρούς ε, ανεξάρτητους επιχειρηματίες είναι πάντοτε οι ίδιοι. Τώρα, σε σχέση με όσα υπόθηκαν από την κυρία Γκογιέν για το δικαιοδότη και το δικαιοχρήστη, εγώ δεν είμαι ειδικό, ε, όμως ε, ε, μπορώ να σας πω ότι αυτός που λαμβάνει τη δικαιοκρισία είναι έχει υποδιοκτησία του τη σύμβαση και αυτή η σύμβαση έχει πραγματική αξία γιατί όπως σας είπα τα χρήματα συνδέονται με την ιδιοκτησία του συμβολέου και όχι με την ιδιοκτησία της μάρκας και θέλω να επιμείνω επίσης στο αυτό το ότι αυτό που κατά την άποψή μας εμποδίζει να ε, δεκτούμε περισσότερους λιανεμπόρους ε, διεθνείς είναι ότι οι περισσότερες από τις αρχές μας δεν έχουν κατανοήσει ότι η έλευση ε, νέων εισερχομένων σε ένα playing field δεν είναι απειλή αλλά ευκαιρία. Όσο περισσότεροι είμαστε στην αγορά λιανική, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταργήσουμε αυτή την ομοθεσία που εισαγάγει διακρίσεις γιατί ο μόνος ε, στόχος ε, αυτής της νομοθεσίας ε, είναι να εμποδίσει τους νέους ερχομένους και να εμποδίσει τον ανταγωνισμό. Κυρία Γκογιάννη, σε ευχαριστώ. Τρία σχόλια. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την εδαφική διάκριση, εμείς σεβόμαστε απόλυτα τις επιλογές των ΜΜΕ να μην πάνε διασυνοριακά γιατί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά αυτό που επικρίνουμε είναι αυτό που και αυτό που βλέπουμε και δοκιμάσαμε είναι το εξή. Εταιρείε που είναι παρούσε σε πολλέ χώρε που έχουν διαφορετικέ πολιτικέ τιμολόγηση και που αρνούνται για τον καταναλωτή να πάει διασυνοριακά. Αυτό έχει να κάνει με κατακαιρματισμό τη αγορά. Ο λόγος ε, του κατακαιρματισμού είναι ένας λόγος να μην φύγουν διασυνοριακά οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι ένας λόγος αυτός, αλλά όχι ο κύριος. Νομίζω το ΦΠΑ είναι ο κύριος λόγος για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Υπήρξε μια πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου που έδειξε ότι πάρα πολύ λίγοι εμπορευόμενοι γνωρίζουν τον κατακαιρματισμό. Έτσι λοιπόν, αν δεν το γνωρίζουν, ε, δεν τους εμποδίζει αυτό. Επίση, συμφωνώ ότι πρέπει οι πληροφορίες να είναι χρήσιμε και δεν πρέπει να παρέχουμε υπερβολικές πληροφορίες στον καταναλωτή. Πρέπει να βρούμε δημιουργικού τρόπους ε, για να φτάνουν οι πληροφορίες στον καταναλωτή με έναν εύκολο τρόπο και εύληπτο τρόπο, όμως ε, το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες επί της ετικέτα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές και μπορώ να αναφερθώ σε ισχυρισμού ή σε άλλου είδου πληροφορίε. Και το τρίτο σχόλιο μου έχει να κάνει με την πρόσβαση στα καινοτόμα προϊόντα. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε το οι καταναλωτές ε, έχουν πρόσβαση ε, στα αγαθά όταν είναι σίγουροι για την ποιότητά τους με το ότι ανοίγουν αγορές στην περίπτωση που τα προϊόντα ε, δεν ε, χαίρουν επαρκή ε, πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θέτουμε νέα προϊόντα στην αγορά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι σέβονται την αρχή τη πρόληψη και δεν θέτουν σε κινδύνο την ασφαλή την υγεία των καταναλωτών. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Μονίκ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπεζοβέν. Αν θέλει να πάρει το λόγο για να αναφερθεί στα θέματα που ακούστηκαν. Ε, είναι εμπνευστή της Έκθεση ο κύριος Μπενζεμάν και ε, έχει επιτελέσει και τη μελέτη για την ε, λιανική αγορά. Έχω δύο ερωτήσεις για το direct selling, τις άμεσες πωλήσει. είναι κάτι που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό τμήμα διαφοροποίηση των πορείων στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρος να συμπεριληφθεί και αυτό στην έκθεση, αλλά πρέπει να διαδραματίσουμε ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασία και φυσικά η γενική επιχειρηματικότητα θα ευνοήσει και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε στον ε, Λονδό συνάδελφο να πω ότι είναι φυσικά οι δικοί σας λιανέμποροι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ε, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά σημεία στα οποία θα αναφερθούμε, τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών και της ελεύθερης δυνατότητας αγοράς σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, κύριε Βεζαμένα, αν έχετε κάποια σχόλια εκ μέρους της Κομισιόν, θέλω να σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς και την Επιτροπή σας που οργανώσατε τη σημερινή συνάντηση που μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πιο πολύ ακούμε σήμερα παρά παίρνουμε θέση. Όσον αφορά τις συζητήσεις που ακούσαμε θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Ε, έχουμε ακούσει αλλού ότι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, είναι αντικείμενο του ε, νόμου περί ανταγωνισμού. Αυτό όμως, ε, με αυτό διαφωνώ, διότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει δεσπόσα θέση στην αγορά και αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες. Υπάρχουν κανόνες στον τομέα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στα περισσότερα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με τον δόκτωρα Ντέιβις ε, που έχει αποχωρήσει ε, ότι δεν είναι δεν αποτελούν πρόβλημα επειδή διαφέρουν μεταξύ τους. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή στον τομέα αυτών. Έχουμε ήδη αρχίσει να εξετάζουμε το θέμα αυτό αναλυτικά. Άλλη παρατήρηση για το θέμα αυτό. Υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο τελευταίες ε, συζητήσεις ε, λόγω, στους, λόγω των ε, Ολλανδών ανεξάρτητων Ελιανοπολιτών. Κάποιες ρήτρες σε συμβάσεις franchising είναι σίγουρα θέμητες και Γι' αυτό επικροτώ την ε, σχετική παρουσίαση που έγινε. Και τέλος, όσον αφορά τα στοιχεία όσον αφορά τον εδαφικό κατακαιρματισμό αυξάνονται. Θα πρέπει να υπερεξετάσουμε τους λόγους. Είναι σαφές όμως ότι και εμείς λαμβάνουμε παράπονα καταναλωτών λόγω του ότι δεν μπορούν να λάβουν τα προϊόντα που έχουν παραγγείλει επιγραμματικά ή ε, τους παραπέμπει στο σελίδα στην δική τους χώρα για να αγοράσουν τα προϊόντα. Η σχετική έκθεση τόνισε σαφώς ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μέρος του λιανικού εμπορίου. Ε, δεν πρέπει να θεωρηθεί τελείω ξεχωριστή δραστηριότητα. Αρκετοί ομιλητέ το ανέφεραν αυτό σήμερα. Τέλο, όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι σαφέ ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες και η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε κάποιο τύπου απλοποίηση, ειδικά στην ε, κατάργηση των οικονομικών ε, δοκιμών, αλλά στην έκθεση για το λιανεμπόριο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα διασυνοριακό πρόβλημα. Το 30% των πολιτών μας ζουν σε ε, περιοχές κοντά στα σύνορα και συχνά περνούν τα σύνορα για να ε, αγοράσουν προϊόντα. Εάν δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα ε, στις αρχές των διαφόρων χωρών, ε, μπορεί να έχουμε στρέβλωση των συνθήκων. Δεν λέμε ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ενιαίο σχέδιο. Θα πρέπει όμως να αναγνωριστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Μια σειρά κρατών μελών εξετάζουν την ε, δημιουργία συστήματος ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για να αποφευθούν ε, τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, η πληροφόρηση των καταναλωτών είναι βασικό θέμα και μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το διαδίκτυο για να βελτιώσει την πληροφόρηση προς τους καταναλωτές. Αλλά η πληροφόρηση θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε περίπτωση επιγραμμικών προσφορών, αλλά και ε, σε περίπτωση διασυνοριακών προσφορών ε, οι καταναλωτές. Ε, κοιτούν τα προϊόντα σε μια ακτίνα διαδρομής 15-20 λεπτών από το μέρος που μένουν. η καλύτερη πληροφόρηση θα βοηθήσει την επιλογή των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πασοφέ. Προχωρούμε στο επόμενο πάνελ μας που έχει να κάνει την, ε, τις ε, βιώσιμες καταναλωτικές ε, συνήθειες. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα. Το θέμα της βιώσιμης κατανάλωσης είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές σε καθημερινή βάση. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μας πείτε ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο ρόλος των λιανοπολιτών στις καταναλωτικές συνήθειες ε, του Ευρωπαίου πολίτη. Πώς μπορεί δηλαδή ο Ευρωπαίος πολίτης ε, να ε, καταναλώνει ενέργεια με βιώσιμο τρόπο και άλλα. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ροντρίγκο Κουβέγια που από την Eurocoop, όλοι την γνωρίζουν θα μας μιλήσει λοιπόν για κάποιες πρακτικές τις οποίες ε, εφαρμόζουν ήδη πολλοί λιανοπολιτές. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό επίσης. Οι λιανοπολιτές ε, ε, ασχολούνται και με θέματα καινοτομία. Αυτό ίσως να μην είναι γνωστό αρκετά. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε περισσότερα από εσά. Πέντε λεπτά έχετε. Thank you very much. Is it Uh, Σας ευχαριστώ για την πρόκληση. Πέντε λεπτά έχω μόνο, Επομένω, θα είμαι τηλεγραφικό. Βλέπετε εδώ τι κουκίδε στα θέματα τα οποία θα αναφερθώ. Να σα πω ότι η Eurocop αποτελεί ένα πολύ σημαντικό είδο ε, λιανεμπόρων. Ε, δημοκρατικά ο έλεγχο γίνεται από του ίδιου των καταναλωτέ. Πρόκειται για καταναλωτικού συνεταιρισμούς. Κυρίω ασχολούμαστε στον τομέα των τροφίμων δραστηριοποιούμαστε στον μέτρο Άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι δραστηριοποιούμαστε στην αγορά σύμφωνα με ορισμένε αξίε ε, και κάποιες αρχές. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ε, αγορά λιανικού εμπορίου και ε, αυτή η συνεισφορά έχει να κάνει με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αηφορία. Καταρχήν, εκεί εισάγουμε τις αρχές μας. Οι αρχές μας έχουν να κάνουν με τη δημοκρατική συμμετοχή των καταναλωτών, την επιρροή που ασκείται επί της διαχείρισης της επιχείρησης από τους καταναλωτές, την ελληνική μεταξύ των γενεών κτλ δεν ε, ζητούμε να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος, αν και επιζητούμε κέρδος, δεν θέλουμε να το μεγιστοποιήσουμε, αλλά ε, θέλουμε να απαντήσουμε στις ανάγκες και στις προσδοκίες των καταναλωτών. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα για το τι κάνετε, ποιοι είναι, γιατί όλοι ξέρουμε ε, ποιοι είστε, αλλά χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία για τη δική μα έκθεση. Θα φτάσω και σε αυτό, λέει ο Ε, Έχουμε μικροπρόθεσμη προοπτική. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, θέλουμε να έχουμε μια εταιρική σχέση με του προμηθευτέ. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά αν ε, υπάρχουν προβλήματα θέλουμε να τα συζητήσουμε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν ε, συνθηκολογούμε, πάντοτε υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θα φτάσω και σε παραδείγματα αμέσως. Ένα από τα κυρία εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την παροχή αυτών των αξιών στους καταναλωτές είναι μέσω των προϊόντων ιδιωτική ετικέτας και ήμασταν στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη προϊόντων όπως είναι προϊόντα χωρίς γενετικά τροπομένους οργανισμούς, βιολογικά προϊόντα με οικολογική ετικέτα και τα λοιπά. Θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, θα σας αναφέρω τι συγκεκριμένα κάνει η Eurocop. Υπάρχει μια συμφωνία με μια οργάνωση ε, που ε, χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία που έχει δημευτεί από τη μαφία προκειμένου να ε, παράξει τρόφιμα συνήθως και αυτά διατίθενται ε, σε όλη την Ιταλία με μια συγκεκριμένη μάρκα. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε εμείς ε, να ε, εισαγάγουμε τη βιωσιμότητα. Ένα ακόμη θέμα που θέλω να τονίσω έχει να κάνει με την ένδειξη των παραγωγών στα προϊόντα μας και στα προϊόντα ίδιας ετικέτας μας. Πολλές φορές ακούγεται κριτική ότι δεν αναφέρονται τα ονόματα των παραγωγών και δεν είναι γνωστή παραγωγή στις ιδιωτικές ετικέτες. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι το πράγμα και οι δικές μας ιδιωτικές ετικέτες αναφέρουν ε, το, το όνομα των παραγωγών και προσπαθούμε ε, σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας να γνωστοποιήσουμε τους παραγωγούς των καταναλωτή γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικός ο σύνδεσμος μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών κυρίως όταν μιλάμε για έναν ε, ε ή για μία μικρομεσαία επιχείρηση. Επίσης, ε, θέλω να σας καλέσω να δείτε την έκθεσή μας για την κλιματική αλλαγή. Είχαμε ένα μακρύ κατάλογο ε, βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται από τα μέλη μας στον τομέα της αηφορίας και εκεί συμπεριλαμβάνεται Εντάξει, ένα από τα outlet της Κόπης στην Ιταλία ε, έχει εγκαταστήσει ηλιακά πάνελ και ε, εκεί παράγεται ενέργεια για να χρησιμοποιείται από τους λιανεμπόρους μας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, η ομάδα των συνεταιρισμών έχει αποθήκες και γραφεία και το 98% της ενέργειας που χρησιμοποιείται εκεί προέρχεται από ενώσιμες πηγές. Αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω, για να κλείσω, τι λένε και οι άλλοι σε σχέση με το συνεταιριστικό μοντέλο. Το 2012 θα είναι το διεθνέ έτο του ΙΕ για του συνεταιρισμού. Τα Ηνωμένα Έθνη γνωρίζουν ότι οι συνεταιρισμοί αναπτύσσουν ε, ένα καλύτερο κόσμο. Υπάρχει μία μελέτη ε, η οποία λέει ότι είναι πιο ανθεκτικό το συμμετεριστικό μοντέλο στην κρίση. Ε, αναπτύσσονται κάποιες ε, πολιτικές ε, που αφορούν τους λιανεμπόρους. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά ξέρω ότι δεν έχω χρόνο. Έτσι λοιπόν, τελικό συμπέρασμα. Θέλουμε να δούμε στην έκθεσή σας την προώθηση του μοντέλου του συνεταιριστικού ως ένα από τους τρόπους για μεγαλύτερη συνοχή και καλύτερη συνδεσιμότητα των πολιτών με την ενιαία αγορά σας. Ευχαριστώ για τις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σας για την έκθεσή μας. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μάτιν Βάιντεστρατ, ο οποίος ε, είναι ε, διευθυντής ε, ευρωπαϊκών υποθέσεων στο IKEA. Σας καλέσαμε γιατί το IKEA είναι στην πρώτη γραμμή ενός μοντέλου που έχει θετηθεί και από πολλούς άλλους εμπόρους λιανικής, κυρίως από τη στραγγυλή τράπεζα των λιανεμπόρων σε ό,τι αφορά την μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε κατευθείαν στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την IKEA. Κύκλος εργοσιών 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράγουμε στην Ευρώπη και έχουμε 127 περίπου χιλιάδες συνεργάτες. Το σημαντικό ζήτημα για μας στην εσωτερική αγορά είναι ο ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έρχονται σε μας και ότι εμεί μπορούμε να του προσφέρουμε προϊόντα χαμηλού κόστου για το σπίτι του, έχοντα μια καλύτερη παραγωγή, καλύτερη λειτουργία τη αλυσίδα εφοδιασμού. Ξέρουμε από διάφορες μελέτες ότι, περί, ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού οδηγεί σε λιγότερη καινοτομία, λιγότερες θέσεις εργασίες, λιγότερες επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και ότι έχουμε λιγότερα προσιτά βιώσιμα προϊόντα για τον καταναλωτή που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το σπίτι του. Πώς μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη, καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανταγωνισμό για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Στο IKEA ξεκινήσαμε με τις επίπεδες συσκευασίε καθώς επίσης και με φύς τρόπους μεταφοράς των προϊόντων. Αυτό το κάναμε αρχικά για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο όμως να κάνουμε και τα προϊόντα λιγότερο ακριβά και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Επίση, χρησιμοποιήσαμε διάφορες ε, μεθόδους ε, από τις ε, εταιρείες που κατασκεύαζαν πόρτες προκειμένου να καταφέρουμε να συσκευάζουμε καλύτερα τα προϊόντα μας και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε με, την, με μικρότερη κατανάλωση καυσίμων. Επίσης, φορτώνουμε τα προϊόντα μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται λιγότερα φορτηγά. Κατά αυτόν τον τρόπο γεμίζουμε περισσότερα κοντέινερ και επιβαρύνουμε περισσότερο, λιγότερο με συγχωρείτε, μέσω των μεταφορών μας το περιβάλλον. Ξέρω ότι πολύ συχνά η εξοικονόμηση χρημάτων και το περιβάλλον συνδέονται και είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο ανταγωνισμού για να αποφελούμε θα και εμείς και οι ανταγωνιστές μας. Τώρα, βιωσιμότητα στο σπίτι, έχοντας μειώσει το κόστος των προϊόντων και έχοντας βελτιώσει τα προϊόντα μας, έχουμε δημιουργήσει και ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τον ίδιο του καταναλωτή. Βλέπετε εδώ πέρα ένα φωτιστικό, το Γιάνσο, το οποίο το έχω φέρει εδώ μαζί μου, να το δείτε και όλοι σας. Έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ θετικό παράδειγμα πώς ε, η αυξημένη παραγωγικότητα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση της τιμής, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να το αγοράσουν και να μειώνεται ουσιαστικά και η κατανάλωση ενέργειας. Αυξήσαμε τις πωλήσει από 300.000 σε 5 εκατομμύρια ετησίως. Χρησιμοποιείται εδώ πέρα ένας μόνο γλόμπες και η κατανάλωση ενέργεια είναι πολύ χαμηλή. Ο ανταγωνισμό είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη καινοτομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ανταγωνισμό να περνάει από το εθνικό στο κοινοτικό επίπεδο και κατά αυτόν τον τρόπο να οδηγεί σε μείωση των τιμών, να οδηγεί σε μεγαλύτερε επενδύσεις, σε καλύτερη βιωσιμότητα. Επίσης θα πρέπει μέσω της καινοτομία να μειωθούν όλα, να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια, τα εμπόδια με συγχωρέ, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εσωτερική αγορά. Με τα εμπόδια αυτά, με την παρουσία των εμποδίων αυτών, θα καταφέραμε να λειτουργήσουμε καλά στην εσωτερική αγορά και θα στρεβλώνονταν ο ανταγωνισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι σε όλα τα επίπεδα τη εσωτερική αγορά ο ανταγωνισμό λειτουργεί σωστά. Σα ευχαριστώ πολύ και είμαι και στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Uh, ευχαριστώ. Ήσασταν σύντομο ο Σουηδό που είστε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ξαβιέχουα που είναι διευθυντής της Efficient Consumer Response και μπορεί να μας εξηγήσει πώς μπορούν οι κατασκευαστές και οι λιανοπολιτές να συνεργαστούν προς όφελος ε, του καταναλωτή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι. Όπως αναφέρατε, το ECR δεν είναι η ε, ομάδα Ευρωπαίων ε, ε, Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Του να είναι, σημαίνει αποτελεσματική αντίδραση των καταναλωτών. Να σας θυμίσω σύντομα την αποστολή μας. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή πλατφόρμα όπου συμμετέχουν λιανοπολιτές και παραγωγοί. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε για να ε, ε, πληρούμε τις επιθυμίες των καταναλωτών ε, καλύτερα, πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος. Έτσι, περνώ στην επόμενη διαφάνεια όπου βλέπετε ένα δίκτυο των οργανώσεων της ECR όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιφερειές του κόσμου επίσης. Υπάρχει το Consumer Goods Forum που είναι ε, διεθνής οργάνωση. Βλέπω ότι οι διαφάνειες περνούν πολύ γρήγορα και δεν προλαβαίνω να τα πω. Η βασική ιδέα της οργάνωσής μας ε, είναι να έχουμε ε, δραστηριότητες ε, σχετικά με την ε, αποτελεσματικότητα μέσω της ε, συνεργασίας καταναλωτών και παραγωγών για να ικανοποιήσουμε τους καταναλωτές. Σας δείχνω εδώ κάποια παραδείγματα από μια μελέτη που έγινε πριν πέντε χρόνια που ισχύει ακόμα όμως. Βλέπετε τη διαφορά ανάμεσα τις, στους λιανοπολιτές και τις, ε, για τους παραγωγούς που έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές της ECR και αυτούς που δεν έχουν υιοθετήσει την, ε, τις πρακτικές της ECR ε, και όπως τα βλέπει ο καταναλωτής. Βλέπετε γενικά ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές της ECR τα πηγαίνουν καλύτερα από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές αυτές. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από τους ίδιους τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, στο, ε, στην τελευταία γραμμή βλέπετε την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ε, στα γράφια των καταστημάτων βλέπετε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει τι πρακτικές της CCR διαθέτουν καλύτερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές αυτές. Επόμενη διαφάνεια. Ένα παράδειγμα του τι έχει κάνει η ECR. Ε, σας δίνω στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ε, στον τομέα των ε, βιώσιμων μεταφορών. Βλέπετε τα στοιχεία που αφορούν τη Γαλλία. 13 επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές και τις διαδικασίες που έχει αναπτύξει η ECR. Πράγμα που επέτρεψε εξοικονόμηση 1.500 τόνων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα Βλέπετε την εξοικονόμηση και σε λίτρα καυσίμων 563-503. Ε, το ίδιο ισχύει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε φορά που η ECR ασχολείται με ένα πρόγραμμα ε, όπως αυτό που αφορά τις ε, βιώσιμες μεταφορές, οι επιχειρήσεις υπολογίζουν το όφελός τους. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα φυσικά, όχι στη διαφάνεια αυτή. Θα σας αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ε, αποβλήτων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και των απορριμμάτων. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Οι επιχειρήσεις που ε, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν του χρόνου να εξοικονομήσουν, μάλλον να αποφύγουν την παραγωγή 75.000 τόνων απορριμμάτων Μιλάμε για πρόληψη δηλαδή και ταυτόχρονα 150.000 τόνοι ε, απορριμμάτων ε, θα ε, δεν θα πάνε στις ε, χωματερές ε, και έτσι θα γλιτώσουμε τον, την προσπάθεια που χρειάζεται για τη διαχείριση των απορριμμάτων αυτών. Νομίζω ότι η συμβολή της ECR στην Εστρογγυλή Τράπεζα ε, οφείλεται στο ότι οι λιανοπολιτές και οι παραγωγοί συνεργάζονται για να πετύχουν καλύτερες λύσεις, να εφαρμόσουν λύσεις οι οποίες τελικά θα, είναι, θα ωφελήσουν τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω και πάλι τον κύριο Χάρμπουρ και να του δώσω το λόγο, να δώσω σε άλλον το λόγο. Θέλει κανείς να προσθεθεί στον κατάλογο των ομιλητών διαφορετικά να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Κίλπεκ από το Σουηδικό Συνδικάτο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη η συμμετοχή μας ε, στην συζήτηση. Ακούσαμε τους διάφορους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο εμπόριο. Ε, αυτό το τμήμα της συζήτησης είχε να κάνει με την βιωσιμότητα και κυρίως ε, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Ε, εγώ πιστεύω ότι σημαντικό είναι όταν μιλάμε για βιωσιμότητα να μιλάμε και για την κοινωνική διάσταση. Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να σκέφτονται και με αυτούς τους όρους όταν, όταν βλέπουν μια μάρκα. Να ξέρουν ότι η μάρκα αυτή αντιπροσωπεύει και ε, κάτι κοινωνικά βιώσιμο. Και γι' αυτό θα ήθελα να συμπεριληφθεί μία πρόταση για τους εργαζομένους, μία παράγραφος ε, ε, εργαζομένους ε, στην έκθεσή σας. Ε, θα θέλαμε να είναι πιο δίκαιο το εμπόριο. Ξέρουμε ότι πολλοί που εργάζονται στο εμπόριο ε, δεν έχουν υψηλή εκπαίδευση, πρέπει όμως να ασχολούνται με θέματα νέων τεχνολογιών και τέτοια. Οι καλές συνθήκες δημιουργούν και ένα αίσθημα ασφάλειας και το αίσθημα ασφάλειας ε, με κάνει καλό υπάλληλο και ε, καλό ε, προωθητή της μάρκας που εκπροσωπώ και αυτό συμβάλλει στην βιωσιμότητα. Έτσι δημιουργείται ένα καλό κλίμα στο χώρο εργασίας. Πολλές ε, σουηδικέ επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν και μια σειρά βασικών αξιών που θέλουμε να προωθήσουμε. Σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να προωθηθούν ε, οι αρχές αυτές άσχετα από την ε, μορφή της επιχείρησης. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις franchising κλπ και για να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε σημαντικό είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για κοινωνικό διάλογο και σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ε, και σε τοπικό επίπεδο. Αυτά ήθελα να προσθέσω. Είναι λοιπόν σημαντικό να συμπεριλάβουμε και την ε, κοινωνική διάσταση όταν μιλάμε για βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ Μαρή. Δίνω τώρα το λόγο και έκλεισε το μικρόφωνο της από την πλατφόρμα βικιλότητας του Βελγίου έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ζούμε λοιπόν για την πλατφόρμα βιοπικιλότητας του Βελκίου. Το Νοέμβριο του 2010 οργανώσαμε μια διαβούλευση 230 Ευρωπαίων πολιτών ε, για θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιοπικιλότητα. Έτσι λοιπόν λάβαμε μια σειρά συστάσεων προς εφαρμογή προκειμένου να αποφύγουμε την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και την απώλεια βιοπικιλότητας. Οι πολίτες μεταξύ άλλων ε, ζήτησαν μεγαλύτερο έλεγχο στην ε, αλυσίδα προμήθεια προκειμένου να αποφευκτούν αθέμητε πρακτικές ή παράνομες πρακτικές και πρότειναν να βελτιωθούν οι ετικέτε, δίνοντας ε, στον καταναλωτή δυνατότητα αξιολόγησης ε, της παραγωγής. Αν παίρνουμε το σχάρι, ε, αγοράζουμε τώρα ένα προϊόν, ε, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για το οικολογικό το αποτύπωμα ή αν αγοράζουμε, παίρνουμε το σχάρι ένα τραπέζι, θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται και πώς κατασκευάστηκε. Έτσι λοιπόν, αυτό ζητείται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι πολίτες επίσης ζήτησαν να γίνουν περισσότερες προσπαθίες για τη μείωση των αποβλήτων ε, με τις συσκευασίες των προϊόντων αλλά και ε, βελτιώνοντας ε, και τι συσκευασίε μέσω τη χρήση λιγότερου πλαστικού, παραδείγματο χάρη. Η έννοια τη βιοπικιλότητα και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων θα πρέπει να αναφέρεται ευρέω στα καταστήματα λιανική. Αλλά ε, επίσης θα πρέπει να αναφέρεται και ένας ε, κωδικός βιωσιμότητας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους λιανεμπόρους για να δείξουν ότι έχουν ε, δεσμευτεί και λαμβάνουν υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποια βήματα προς τα μπρος ό,τι αφορά την ενέργεια, το είδωρ κτλ. Σήμερα όμως δεν περιλαμβάνονται η βιοπικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ στη δική μας πλατφόρμα να παράσχει κάποιες προτάσεις και η ιστοσελίδα μας αποτελεί και μια πλατφόρμα πολιτών για να συζητήσουν με όσους αποφασίζουν και χαράσουν την πολιτική. Θέλουμε λοιπόν να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτήν την πλατφόρμα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπέχο, τώρα κυρία Ελάρια Σαβοίνη, η οποία είναι σύμβουλος κοινωνικών υποθέσεων στο Commerce. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Κορατσαμπίλτ, πολύ σύντομη θα είμαι, ούτε καν δύο λεπτά δεν θα μιλήσω. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πτυχές που γνωρίζετε και είναι σημαντικές για τους κοινωνικούς εταίρους του εμπορικού τομέα και που ήδη αποτέλεσαν αντικείμενο της κοινή θέση. Πρόκειται για γενικά θέματα, τα οποία δεν συνδέονται μόνο με κοινωνικά αλλά και οικονομικά ζητήματα προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία του τομέα του λιανεμπορίου. Θεωρούμε σημαντικά δύο θέματα. Καταρχήν την καταπολέμηση της παραοικονομίας και δεύτερο να εργαστούμε από κοινού για να βελτιώσουμε το συντέριασμα ε, των αναγκαιοτήτων ε, των επιχειρήσεων ε, για δεξιότητες και των προσόντων που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει και μία ανακοίνωση για το θέμα της απασχόλησης και υπάρχει μια πλατφόρμα για τα κοινωνικά ζητήματα η οποία λειτουργεί πολύ καλά. Και τέλος, ο κύριος Χάρμπουρ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, ένα Μαρία. Και εγώ έχω δύο λεπτά όπως όλοι άλλοι. Μια σκέψη θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. που ουσιαστικά συνδυάζει τα δύο τελευταία πάνελ. Το ζήτημα της οικονομίας κλίμακος, της αποτελεσματικότητας, αλλά και του δυναμικού χαρακτήρα του τομέα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Βίλκεμ και η κυρία Χουγκστράντετ μίλησαν για την σημασία που έχουν οι ανεξάρτητοι λιανοπολιτές και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη και στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Μέρος των ε, ζητημάτων που συζητήσαμε για την αύξηση δηλαδή της αποτελεσματικότητας και για την πιο φιλική προς το περιβάλλον ε, ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου έχουν να κάνουν σαφώς με την ε, ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών αλλά και με τη λειτουργία παράλληλων συστημάτων όπως κοινά συστήματα μεταφοράς προϊόντων και σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα στον τομέα των μικρολιανοπολιτών ή στις μικρές αλυσίδες εφοδιασμού. Στη δική μου ε, περιοχή, για παράδειγμα, υπάρχουν παραγωγοί τροφίμων οι οποίοι διαχειρίζονται το δικό τους μικρό σύστημα μεταφοράς και εφοδιασμού των προϊόντων τους. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται γιατί πολύ συχνά οι μικροί λιανοπολιτές δεν έχουν ε, ε, τα συστήματα εκείνα που θα του επέτρεπαν να λειτουργήσουν όπω οι μεγάλοι λιανοπολιτέ. Δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια συστήματα. Σίγουρα θα μπορούσε η ECR να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε περισσότερο με τους μικρούς λενοπολιτές και προμηθευτές και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε περισσότερο τους, μικρού, τους ανεξάρτητους να συνεργαστούν μεταξύ τους και να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερα συστήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρήσουν αν θέλετε την ανεξαρτησία τους και την ιδιοκτησία τους αλλά έχουν και πρόσβαση σε συστήματα τα οποία λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Και πρέπει να δούμε εδώ πέρα ποιο μοντέλο τελικά θα ακολουθήσουμε. Ένα ανταγωνιστικό μοντέλο ή κάποιο άλλο. Δυστυχώ ο Πίτερ Ντέβι έχει φύγει αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν όλο και μεγαλύτερε εταιρείε, μεγαλύτεροι ελληνοπολιτέ, οι οποίοι προσπαθούν να να μπουν περισσότερο μέσα στον κόσμο των λιανοπολιτών και να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους μικρά δίκτυα πρόθεση των προϊόντων. Θα είναι πρόβλημα, αυτό είναι κάτι θετικό. Σας ευχαριστούμε Μάλκομ. Ολοκληρώνουμε δίνοντα το λόγο στου ομιλητέ μας. Ο κύριος Ροντρίγκο Γκουβέα, πρώτος από την ε, Eurocop, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Α μιλήσουμε για το ζήτημα της κοινωνικής βιωσιμότητα, στο οποίο αναφερθήκαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική βιωσιμότητα. Έχουμε ήδη κάποιε βέλτιστες πρακτικέ στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ε, πρότεινα να διαβάσετε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών και θα δείτε ότι ε, η ΚΟΠ στην Ιταλία και η ΚΟΠ στην Δανία είναι οι ε, δύο μεγάλες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν θετική βαθμολογία όσον αφορά την κοινωνική βιωσιμότητα. Επίσης, τα μέλη μας έχουν ένα κώδικα διντολογίας όσον αφορά την σήμαση των προϊόντων όσον αφορά την εισαγωγή των προϊόντων ε, από τρίτες χώρες, κυρίως από χώρες της ε, Νότια-Ανατολικής Ασίας και ο κώδικας αυτός δολογίες αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα όπως η παιδική εργασία ή τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Μπορώ να σας δώσω λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης εργαζόμαστε πάρα πολύ για το fair trade, το δίκαιο εμπόριο, το γεγονός ότι ε, το ζήτημα αυτό αφορά ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι θετικό. Υπάρχει μια ομάδα εργασία στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τώρα του τους μεγάλη κλίμακα κλίμακας και τους μικρούς λενοπολιτέ, του ανεξάρτητους. Αυτό το οποίο μπορούν να εγγυηθούν οι συνεταιρισμοί είναι ότι έχουμε κάποιες μικρές εταιρείες, 3.500 συγκεκριμένα, την ιδιοκτησία των οποίων έχουν άνθρωποι από την ίδια περιοχή, επομένως η ιδιοκτησία βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο και τα κέρδη από τις εργασίες των εταιριών αυτών επιστρέφουν πίσω στην τοπική αυτή κοινότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το σύστημα αυτό. Ο συνεταιριστικός τρόπος εργασίας επικεντρώνεται πάρα πολύ στο τοπικό στοιχείο, στο τοπικό παράγοντα. Σκεφτόμαστε τοπικά, εργαζόμαστε τοπικά και τα κέρδη επιστρέφουν στον, στον ίδιο τόπο. Πρόεδρος. Σίγουρα θα δούμε τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στην έκθεση αυτή, τέσσερις σελίδες συγκεκριμένα. Μάρτιν, έχετε το... Μπορείς να μιλήσεις για δύο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι κάπως ε, δύσκολο να συνοψίσω το τι κάνουμε στην IKEA και όσον αφορά την κοινωνική διάσταση και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Έχουμε μια σειρά προγραμμάτων και εδώ στην Ευρώπη και στην Ινδία. Στην Ινδία, για παράδειγμα, 80.000 βαμβακό παραγωγή 80.000 βαμβακοπαραγωγούς βοηθούμε να αναπτύξουν τα συστήματά τους. Ε, πολλά παιδιά αποφαλούνται στα σχολεία τους από τα προγράμματα μας. Ε, ήθελα να τονίσω όμως ε, το θέμα του ανταγωνισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό είναι να μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε ανταγωνιστικά μεταξύ μας, να μπορούμε να ε, έχουμε καινοτομία, να υπάρχει κάποιος που να μας ε, στηρίζει, που να, ε, βοηθάει, που να εργάζεται και προς όφελος του μικρού λιανο, λιανέμπορου και του μεγάλου. Αυτή η λάμπα εδώ μπορεί, σας δείχνει για παράδειγμα πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο. Όπως και να γυρίσουμε το θέμα, τελικά ο ανταγωνισμός ε, είναι ε, η κινητήρια δύναμη της ε, εσωτερικής αγοράς και της καινοτομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ξαβιαϊουά. Από το ECR για δύο λεπτά. Θα βασιστώ, είπε ο κύριος Χάρμπορ. Το ECR ε, θέλει να απαντήσει στις ανάγκες των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Ε, οικοδομούμε τώρα μια εταιρική σχέση στη Γαλλία. Μεταξύ του ECR ε, Γαλλίας και της Ομοσπονδίας Μικρών και Μεσών Επιχειρήσεων της Γαλλίας και στο, στο Tour de France ε, έχουμε ε, χρησιμοποιήσει κοινέ ε, αποθήκες και μεταφορά θέλουμε λοιπόν να διαδώσουμε αυτή την πρακτική. Αλλά γιατί είναι σημαντικό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις να μοιραστούν τους τρόπους μεταφοράς με τους εταίρους τους στην περιφερειά τους, σε περιοχές όπως τη Βρετάνη ε, πρέπει να υπάρχει επιμερισμός των πόρων ε, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν να εμπορεί. Και κάτι ακόμη που θέλω να αναφέρω για τα θέματα βιωσιμότητας. Η ECR ε, Ευρώπη είναι επίσης το ευρωπαϊκό σκέλος του Consumer Goods Forum και αυτό το φόρουμ ε, πρόσφατα εξέδωσε δύο ψηφίσματα, ένα σε σχέση με την ψήξη και ένα σε σχέση με την αποψήλωση των δασών. Και η ECR Europe θα λάβει αυτά τα δύο ψηφίσματα και θα τα παρουσιάσει ε, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στις ευρωπαϊκές χώρες ε, προκειμένου να τις υποστηρίξει και για να δούμε σε επίπεδο χώρας ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση για την αποψήλωση. Ένα παράδειγμα, το αναφέρει και ο Μάρτιν, η χρήση των παλέτων ξύλου. Υπάρχει εναλλακτική. έτσι λοιπόν ερευνάται στη Γαλλία η χρήση σύνθετων ινών παραδείγματο χάρη αντί να χρησιμοποιούμε ξύλο. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να ολοκληρώσω και αυτή την, αυτό το τμήμα της συνεδρίασης για την εφόρο κατανάλωση. Πολύ σημαντικό. Δεν θα είναι κεντρικό τμήμα της έκθεσης μου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να ζητήσω από εσά του ε, προμηθευτέ, του λιανεμπόρους, του καταναλωτέ του εργαζομένου, να ενώσετε την, ε, δυνάμει σα για να καταπολεμήσουμε τη δημιουργία αποβλήτων. Αυτό έχει οικονομικές ε, και περιβαλλοντικές πτυχές αλλά και άλλες πτυχές. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να κλείσω τη συνεδρίαση λέγοντας καταρχήν ότι για μένα ως εισηγήτρια και είμαι σίγουρη ότι και κάποιοι ε, συνάδελφοι θα συμφωνήσουν. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να σας ακούσουμε και χαρήκαμε πάρα πολύ. Ε, ήταν ε, πραγματικά πολύ δυναμική η ανταλλαγή. Δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχε και τέτοια αντιπαράθεση μεταξύ ορισμένων ξημών και είναι πάρα πολύ υγιές αυτό. Ε, σήμερα τι προκύπτει από τη συζήτηση μία βούληση ε, που εκφράστηκε από τα μέλη των οργανώσεων να ξεκινήσουν και να συμμετέχουν σε ένα διάλογο που να βασίζεται ε, όχι στη θεωρία αλλά σε δεδομένα και προκειμένου να παρουσιάσουμε επικοδομητικέ λύσει προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ τις διάφορες οργανώσεις, το Eurocorona την ΕΤΗ ε, και άλλους όσου εκπροσωπηθήκαν εδώ σήμερα. Ελπίζω στο μέλλον να συμμετέχουν και άλλε οργανώσει και φυσικά ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Τώρα, ε, εσείς μας καλέσατε για το να αποκτηθεί περαιτέρω ορμή στην ελληνική αγορά. Θέλετε να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογή από τα αγαθά στις υπηρεσίες. Ε, θεωρείτε ότι οι ανέμποροι προσφέρουν και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Ε, θέλετε να αναγνωριστεί ο ρόλος των ανέμπορων για το ότι διατηρούν χαμηλό τον πληθωρισμό. Και επίσης ε, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις εις βάρος ποιου ε, δημιουργούνται, μάλλον ε, υπάρχουν αυτές οι χαμηλές τιμές. Και ε, τελικά πώς γίνονται οι επιλογές των καταναλωτών. Υπάρχει μια ξεκάθαρη έκκληση για εναρμόνιση και για σεβασμό της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να αποφύγονται τα διτά πρότυπα, οι διτές ερμηνείες και οι διπλές δοκιμές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρατε και περιμένουμε και άλλα. Ε, αναφερθήκατε σε εμπόδια, στην αγαθά και στις αναφερθήκατε στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα 500 εκατομμύρια καταναλωτών στα 27 κράτη-μέλη σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην ε, Νοτιοκεντρική Ευρώπη. Αναφερθήκατε στο θέμα του φόβου και ανησυχίας που υπάρχει στην αλυσίδα των προμηθευτών και αυτό δεν πρέπει να το αρνηθούμε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επικοδομητικά. Υπάρχει ανάγκη να ανοικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην ε, αλυσίδα προμηθειών και τι θα μπορέσουμε εμείς να βάλουμε στην έκθεση ε, ενίσχυση και εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας πίσω στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν διδεσμοί μέτρων για τα αγαθά και την ε, οδηγία για τις επιχειρήσεις ε, να καλέσουμε την Κομισιόν να διαδραματίσει το ρόλο της ως εποπτική αρχή άρση των υλικών εμποδίων στα οποία αναφερθήκατε σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της εγκατάστασης. Ε, δεν αποκλείω ότι θα υπάρχει και έκκληση ε, στην Κομισιόν για διαδικασίες επί και μπορεί να βρούμε και τρόπους επιτάχυνσης ε, αυτών των διαδικασιών επί παραβάση και φυσικά θέλουμε να εφαρμόσετε πλήρως ε, και η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, το δίκαιο του ανταγωνισμού. Υπήρξαν και κάποιες εκκλήσεις για περισσότερη νομοθεσία, άλλες εκκλήσεις για αυτορύθμιση, για λιγότερη νομοθεσία, για εκούσια μέτρα. Άλλοι είπαν ε, ότι οι κώδικες δεν λειτουργούν, άλλοι είπαν θέλω περισσότερους κώδικες και ε, άλλοι είπαν πρέπει να κάνω μια πολιτική συζήτηση στο επιμελητήριο για το ε, αξιολογήσουμε. Η Κομισιόν είπε ότι δεν αρκεί ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, άλλοι είπαν το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν ε, και διαφορετικές αποκλίνουσες απόψεις από τους ανεξάρτητους φορείς και ανυπομονούμε να εργαστούμε πιο στενά με την Κομισιόν για να δούμε με πιο καλύτερο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των συμβατικών σχέσεων. Για την αηφορία ακούσουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα από τον κλάδο. Είναι πραγματικά ευπρόσδεκτα, σας ενθαρρύνουμε και θα είμαστε θετικοί στην έκθεση για το θέμα αυτό. Τώρα, σα αναφέρω το χρονοδιάγραμμα, συνεχίζεται το διάλογος αυτό ελπίζω. Το μόνο που δεν έχουμε είναι χρόνο, αλλά έχουμε βούληση να σα ακούσουμε, να συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί σα. Υπάρχει βούληση αυτή, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Εσωτερική Αγορά το Φεβρουάριο. Η προθεσμία για μένα παρουσιάσω την έκθεση είναι η Δευτέρα Μαρτίου. Κατόπιν θα έχουμε μία συζήτηση στην ε, Επιτροπή ΙΜΚΟ 21 και 22 Μαρτίου τροπολογίες μέχρι τις 24 Μαρτίου και κατόπιν θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ 13 Απριλίου και στην Ολομέλεια το Μάιο στο Στρασβούργο. Και ελπίζω να είμαι σε θέση να σεβαστώ αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστώ ε, που με εμπιστεύτηκες και την Προεδρία Μάλκο και φυσικά θα είμαστε σε επικοινωνία. Well, Anna um, Άννα Μαρία, θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων, γιατί πραγματικά επινόησες και διοργάνωσες το project αυτό, κατάφερες να προσκαλέσεις τους πάντες. Δεν είναι εδώ πέρα όλοι οι σκιώδεις βέβαια που σε βοήθησαν, αποτελούν όμως και αυτοί πολύ σημαντικό μέρος της όλης συζήτησης. Ξέρω ότι είσαι η συγγήτρια η οποία ακούς πολύ προσεκτικά τους συνομιλητές σου και όλοι ακούσαμε πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα. Πρέπει τώρα να καταφέρουμε να τροφοδοτήσουμε την έκθεσή σου με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή η έκθεση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί μας. Το βασικό μήνυμα της συνεδρίας αυτής που το είπες και πριν από λίγο είναι ότι δεν ξέρω αν καταφέραμε να καλύψουμε όλο τον λιανοπολικό, λιανοπολικό κλάδο, τον κλάδο λιανικής πώληση ή πώς θα καταφέρουμε τελικά να βελτιώσουμε το σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Πάντως σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι όλες οι οργανώσεις που ήρθαν σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουν θα παραμείνουν σε επαφή μαζί μας. Γιατί αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, έναν ενδυναμωμένο διάλογο. Πιστεύω επίσης ότι ορισμένα από τα πράγματα τα οποία γίνονται όπως η ανταλλαγή των πρακτικών, οι συνεταιρισμοί καταναλωτών, οι πρακτικές αυτές οι οποίες δεν βαίνουν κατά του ανταγωνισμού αλλά είναι επωφελείς για τους καταναλωτές, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι υποφελή και για άλλους τομείς πολιτικής πέρα από αυτόν τον οποίο εξετάζουμε. Επομένως, Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση σημερινής συνάντησης θα γίνει και μία άλλη θα συνεδρία για τα μέλη της Επιτροπής μας αύριο σε 9 το πρωί.